Um, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Έχει σχεδόν περάσει ένα τέταρτο από τις τρεις, οπότε προτιμώ να ξεκινήσουμε. Όσοι με ξέρετε, ονομάζομαι Μέρι Χάνη, πολύ με από τις αντιπροέδρους της Επιτροπής των Γυναικών και αντικαθιστώ την ε, ε, πρόεδρό μας, τη Λίνια που έχει πρόβλημα με την πτήση της εξαιτίας του κυκλώνα ε, ζητά συγγνώμη, δυστυχώς όμως ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ακρόση για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα που είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, κατά των γυναικείων καρκίνων. Το Σεπτέμβριο του 2016 οι συντονιστές αποφάσισαν να οργανώσουν αυτή την δημόσια ακρόβαση για να συμπληρώσουν την προγραμματισμένη έκθεση πρωτοβουλίας με τον ίδιο τίτλο και αποφασίστηκε να ανατεθεί έκθεση στην ομάδα EFTD που όρισε την κυρία Γιούτο ως ε, εισηγήτρια. Μία σύντομη εισαγωγή τώρα από μένα. Ε, μία στις τρεις Ευρωπαίες αναπτύσσουν καρκίνο στη διάρκεια της ζωής τους, ε, κάτι που φυσικά δημιουργεί τεράστια προσωπική τραγωδία και οδύνη, αλλά και τεράστιο κόστος για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες μορφές καρκίνου όπως είναι καρκίνος της μήτρας, το τραχύλο της μήτρας και άλλοι καρκίνοι του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, ε, εντοπίζονται κυρίως ε, ε, αποκλειστικά μερικές φορές στις γυναίκες. Παρόλο που αυτές οι μορφές καρκίνου δεν λαμβάνουν τις διάσταση προσοχής ούτε από το ευρύ ούτε από τους ηθήνοντες της πολιτικής. Γι' αυτό με την ακρόασή μας θέλουμε να κάνουμε ένα απολογισμό της παρούσας κατάστασης την πρόληψη, τον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη θεραπεία των γυναικείων καρκίνων και να δούμε τις ε, στρατηγικές που υπάρχουν ή τι χρειάζεται ε, για αυτό το, κλάδο. Οι καλεσμένες μας ε, εμπειρογνώμονες είναι η κυρία Καρεμπέν που είναι αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Europa παντωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το καρκίνο και εκείνη δυστυχώς ε, έχει πρόβλημα γιατί κυρώθηκε η πτήση τη και ε, την δική της παρουσίαση ε, θα την κάνει η κυρία Γιάρετ μετά τη δική της. Τώρα θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Αγιούτου για να μας κάνει την εισαγωγή του θέματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα σε, όλες, σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην ακρόαση αυτή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις εμπειρογνωμονές μας και εκείνες που είναι εδώ αλλά και εκείνες που για λόγους πρακτικούς δεν μπόρεσαν να έρθουν ε, και θα μεριμνήσουν να παρουσιαστεί με τρόπο διαφορετικό η ομιλία τους. Πριν από τέσσερα χρόνια λοιπόν ένας επανερχόμενος καρκίνος του μαστού στήρισε τη ζωή σε μια πολύ αγαπημένη μου νέα μητέρα. Το θέμα λοιπόν που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα με αγγίζει από πολύ κοντά και θέλουμε και να γύρουμε τις συνειδήσεις αλλά και να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών στις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις και να βοηθήσουμε έτσι στην καταπολέμηση αυτού του κακού που όταν ε, πλήττει εμάς τις γυναίκες έχει πολύ σημαντικές και ψυχολογικές διαστάσεις που ε, δεν αξιολογούνται στο απαραίτητο μέγεθος. Είναι διάφοροι οι παράγοντες. Με βάση τα δεδομένα της Eurostat, 600.000 γυναίκες σε όλη την Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους από κάποια μορφή όγκο. Από αυτές, οι 90.000 περίπου ε, πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού. Πρόκειται για εντυπωσιακά στοιχεία. Αλλά είναι πολύ περισσότερες εκείνες οι οποίες ευτυχώς μπορούν να καταπολεμήσουν την αρρώστια, γιατί πάνω από 80% των γυναικών που εμφανίζουν παραδείγματι όγκο στο μαστό μπορούν να ε, επιβιώσουν και σε αυτές πρέπει να απευθυνθούμε μεταξύ άλλων γιατί αλλάζει η ζωή τους κατά τρόπο ριζικό και μερικές φορές και οι συνέπειες μιας χειρουργικής επέμβασης μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικές ψυχολογικές συνέπειες. Επί παραδείγματι μια ιστερεκτομή, μια μαστεκτομή μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες και ψυχολογικό τραύμα σαν συνέπεια που δεν επιτρέπουν ε, να ξαναγυρίσει κανείς το παλιό του εαυτό. Ε, στην έκθεση αυτή που έχω αναλάβει θέλω να υπογραμμίσω όλα αυτά τα ζητήματα και τους προβληματισμούς που σας περιέγραψα προκειμένου τα κράτη-μέλη και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κληθούν να αναπτύξουν πολιτικές και προγράμματα σε θέματα δημόσιας υγείας που θα λαμβάνουν υπόψη ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα προβλημάτων που προκύπτουν από, αυτό το φοβερό, από αυτή τη φοβερή αρρώστια όταν ε, αγγίζει τις γυναίκες. Και στη δική μας την Επιτροπή, με την έκθεση πρωτοβουλίας βεβαίως, ε, αναζητώ και βρίσκω υποστήριξη πολύ σημαντική από τους συναδέλφους, από τις συναδέλφους, πράγμα το οποίο τιμά ολόκληρη την Επιτροπή μας. Σκοπεύω λοιπόν στην πρότασή μου ιδιαίτερα να υπογραμμίσω τρεις βασικές πτυχές. Καταρχάς την πρόληψη παρακολούθηση και πρόσβαση στις αγωγές. Γιατί εραμφίβολα, αμφιβολά η υψηλή συχνότητα της θνησιμότητας που απορρέει από τον ε, όγκο πολλές φορές εμφανίζεται σε μια φάση αρκετά εξελιγμένη της αρρώστιας που δεν επιτρέπει τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη η πρόληψη με μια σταθερή και προσβάσιμη και σε όρους οικονομικούς διάγνωση με γενικές αλλά και ε, ειδικέ εξετάσεις διαγνωστικές. Δεν είναι εύκολο βέβαια να δώσει κανείς απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα όταν ε, οι επισκέψεις ε, για τον έλεγχο το, της υγείας πολλές φορές σημαίνουν και σημαντικά οικονομικά έξοδα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε απαντήσεις. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα για όλες τις γυναίκες σε μια ελάχιστη διαγνωστική ε, και προληπτική διαδικασία και αποτελέσματα σε ε, λογικούς ε, χρόνους. Και επίσης εφόσον υπάρχει πρόβλημα αρρώστιας πρέπει να δίνονται και οι κατάλληλες αγωγές. Πολλές φορές αυτές οι αρρώστιες με τα όργανα τα οποία προσβάλλουν καταστρέφουν την ίδια την έννοια της η, η στη γυναίκα. Και βέβαια η τελευταία πτυχή οικονομική και κοινωνική που σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί υποστήριξη αρρωγή, κατάλληλη για τις γυναίκες που θα περιλαμβάνει κάθε πτυχή μεταξύ των οποίων βέβαια και τις ψυχολογικές ε, συνέπειες, καθώς ε, η ασθένεια πολλές φορές καταστρέφει την ίδια την θηλυκότητα της γυναίκας, τη δυνατότητα της δηλαδή να αισθάνεται ως γυναίκα. Η ψυχολογική υποστήριξη και στην περίοδο που θα ακολουθήσει την αγωγή ή τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει μορφές ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ε, και αρρωγής ε, για κάθε πτυχή της ζωής. Δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν αυτές οι γυναίκες στη μοίρα τους, γιατί η επάνωδο στο ρόλο της μητέρας, της συζύγου, γίνεται μετά την αρρώστια πολύ δύσκολη. Και πρέπει αυτό να το υποστηρίξουμε. Πρέπει λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο τις παρεμβάσεις των εξαίρετων προσκεκλημένων μας που θα μιλήσουν εις βάθος για το πρόβλημα και θα ήθελα να αφήσω το λόγο σε αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιούτο, κυρία Συγγήτρια. Πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εισαγωγή που μας κάνατε. Περνάμε τώρα στις καλεσμένες μας. Η πρώτη εμπειρογνώμη είναι η κυρία Αλεσάνδρα Καμπιτέλη, ψυχολόγος και συνεργάτης πολλών οργανώσεων που παρέχουν ψυχολογική στήριξη. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλεσάνδρα Καμπιτέλη, είμαι ψυχολόγος. Ασχολούμαι με την ε, παροχή υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν εμφανίσει νεοπλασία, αλλά και στις οικογένειές τους. Και στην παρουσίασή μου σήμερα θα ήθελα να σταθώ στις ψυχολογικές πτυχές ε, της ε, αρρώστιας ε, για τη γυναίκα αλλά και για την καθημερινή της ζωή και πάνω απ' όλα την οικογένεια, τη σχέση με τα παιδιά. Αυτό το καθημερινό βίο που κατά κάποιο τρόπο ανατρέπεται, καταστρέφεται, είναι ένα θύμα της ίδιας αρρώστιας. Ο καρκίνος λοιπόν είναι μια πολυσυστημική παθολογία εμφανίζεται και στα κύτταρα και στην ψυχή. Και στα χημικά δηλαδή μόρια, αλλά και στην, στα συναισθήματα. Μερικές φορές βλέπουμε μια, ένα μεγάλο κενό να εμφανίζεται. Όταν αρρωσταίνει από καρκίνο μια γυναίκα, χάνει και την υγεία της αλλά και το σύνολο της ζωής της και τη δυνατότητα για συνέχιση της καθημερινής της και οικογενειακής της ζωής. Όταν μιλούμε για καρκίνο, πάντα έχουμε μια αρνητική εικόνα, μια αρνητική αίσθηση, με πολύ ε, φρικτές εικόνες που έρχονται στο μυαλό που σχετίζονται με την ε, τραυματική εμπειρία της ανακάλυψης αυτής της παθολογίας αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου ζωής πρέπει να γίνουν δεκτές και αγωγές πολύ παρεμβατικές που μπορεί να επηρεάζουν την καθημερινή και φυσιολογική ζωή ακόμη και όταν έχει καταπολεμηθεί η αρρώστια. Ο καρκίνος του μαστού καρκίνος ο οποίος πλήττει ε, μέρος των αναπαραγωγικού συστήματος αλλά ταυτόχρονα και σύμβολο της θηλυκότητας είναι ένας καρκίνος ο οποίος επηρεάζει το ίδιο το σώμα της γυναίκας και της επαναπροσδιορίζει και επηρεάζει την ταυτότητα μέσα στην οικογένεια, τη σχέση με τον σύντροφο, την κοινωνική ζωή λόγω και των φυσικών συνεπειών, των σωματικών συνεπειών των επεμβάσεων στο σώμα, αλλά και περαιτέρω το, τις εμπειρίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να σταθεί και να τις επεξεργαστεί η γυναίκα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να δώσουμε μία ε, υποστήριξη στην διαχείριση αυτής της ογκολογικής αρρώστιας σε σχέση με την εξασφάλιση της ισορροπίας της γυναίκας και της ψυχικής αλλά και σωματικής ισορροπίας. Ωστόσο δεν είναι πάντα δυνατόν να βρεθούν τέτοιες ε, μέθοδοι υποστήριξης ή εάν υπάρχουν αυτές έχουν ε, μια δίσκαπτη δομή και διαχείριση που δεν προσαρμόζονται πάντα στις ανάγκες των ασθενών μας οι οποίες καλούνται να δείξουν ευθύνη και να αναγνωρίσουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να τους προσφέρει τη βοήθεια ή να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται τη ψυχολογική βοήθεια. Πολλές φορές όμως αυτή η ψυχολογική επέμβαση δεν θεωρείται από τις ίδιες ασθενείς ε, απολύτως απαραίτητη, κατεπηγόντως απαραίτητη, ούτε μπορεί να, και επιπλέον μπορεί να μην έχουν τα μέσα για να, την, για να καλύψουν τα εξοδά τη. Πολλέ είναι οι ασθενείς και από πολλέ μελέτε που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία έτη, μπορώ να το πω αυτό, μας λένε ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για την ε, αρρώστια, που τις έχει προσβάλει, έτσι ώστε να λάβουν αποφάσεις για τις αγωγές, τις οποίες ε, μπορεί να αποφασίσουν να υποβληθούν οι μη. Και ακόμη και όταν, οι υπηρεσίες, όταν υπάρχουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, οι ασθενείς αγνούν την ύπαρξή τους την ίδια, τη διαθεσιμότητά τους. Με συνέπειες ε, πολύ σοβαρές για τις ε, πιο ευάλωτες ασθενείς, εκείνες που δεν έχουν μεγάλη, υψηλή κατάρτιση οικονομικά μέσα. Και έτσι επιμένουμε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ισότιμη ε, δυνατότητα πρόσβασης, ισότιμες ευκαιρίες σε αυτή την υποστήριξη. Ε, κάθε χρόνο στην Ευρώπη 150.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου του μαστού εμφανίζονται. Πρόκειται για μια αρρώστια που έχει ψυχική ψυχολογικές εκτός από σωματικές συνέπειες ε, επηρεάζει την καθημερινή ζωή της γυναίκας, την οικογενειακή ζωή, το επαγγελματικό βίο. Τι σημαίνει λοιπόν μια διάγνωση καρκίνου στο μαστό ή άλλου γυναικολογικού καρκίνου στη γυναίκα. Η μαστεκτομή, η, η αφαίρεση των οθικών έχει σημαντικές διαστάσεις ως προς την ε, αντίληψη της θηλυκότητας και του γυναικείου σώματος. Απαιτεί βέβαια την αποκατάσταση του μαστού, πράγμα το οποίο έχει να κάνει με την ε, αντίληψη της γυναίκας για το σώμα της. Πρόκειται όμως πάνω απ' όλα για μια παρέμβαση στη ζωή, στο ψυχισμό, στην ιδέα για το σώμα, στην αυτοεκτίμηση και την αποδοχή της γυναίκας. Βλέπουμε πολλές φορές να εκδηλώνονται και δυσκολίες ε, συναισθηματικού χαρακτήρα. Αισθάνεται η γυναίκα δηλαδή ότι δεν είναι κύριος του ίδιου της του σώματος και δεν μπορεί να ε, ζήσει με τρόπο ομαλό τη σχέση με το σώμα της ή τις ε, σεξουαλικές ε, επαφές. από τις 303 ε, γυναίκες με όγκο σε, στάδιο, σε πρώτο στάδιο και 200 ε, σε πιο προχωρημένο στάδιο καταγράφουν σε 45% προβλήματα ψυχολογικά και ψυχιατρικά για την πρώτη ομάδα και 42% για τη δεύτερη. 36,7% συγκεκριμένα παρουσιάζουν διαταραχές της διάθεσης, 9,6% ε, ελαφραία κατάθλιψη 9% ε, ε, βαριά κατάθλιψη, 27% ε, ελαφρά κατάθλιψη και 8,6% προβλήματα άγχους και, από το... και αντίστοιχα είναι τα δεδομένα και για, το δεύτερο, για τη δεύτερη ομάδα. Ο στόχος λοιπόν που θα πρέπει να επιδιώξουμε θα πρέπει να εξασφαλιστούν, θα πρέπει να εξασφαλιστούν μέσα και για την αγωγή, για τη θεραπεία, αλλά πάνω απ' όλα να μην αισθάνεται η γυναίκα ότι είναι στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της αγωγής. Μια από τις στρατηγικές που θα μπορούσε να υιοθετηθεί θα ήταν η εξασφάλιση καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των γυναικών που έχουν εκτεθεί ε, είτε στην αγωγή ε, είτε στον κίνδυνο του, του καρκίνου και πιστεύουμε ότι έχουν γίνει και αυτό μας το λένε μελέτες που έχουν γίνει ότι όταν υπάρχει ενημέρωση και υποστήριξη από τον ευρύτερο κύκλο η δυνατότητα για ε, αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού, έχουμε μείωση του ποσοστού των ε, εκδηλώσεων άγχους ή ε, κατάθλιψη σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Ωστόσο αυτή η περίθαλψη δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη γυναίκα που έχει εκδηλώσει ήδη τον καρκίνο, θα πρέπει να επεκταθεί στα παιδιά, την ευρύτερη οικογένεια, στο ρόλο της γυναίκας δηλαδή και ως μητέρα, αλλά και ως συζύγου ή συντρόφου. Βλέπουμε μια θετική ε, σχέση ως προς την ε, ε, μια ευθεία αναλογία σε σχέση με την κατάθλιψη ή το άγχος της μητέρας γυναίκας που έχει εμφανίσει καρκίνο και σε αυτήν των παιδιών. Βλέπουμε δηλαδή να αντανακλάται το άγχος και ε, η ψυχολογική πίεση στη γυναίκα και στα παιδιά της. Ο κίνδυνος, ε, ο φόβος της εγκατάλειψης της αρρώστιας της ε, απώλειας στα παιδιά μπορεί να μειωθεί με την ενημέρωση και την ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρεται και στη μητέρα. Έτσι λοιπόν η οικογένεια και για, τον ασθενή, αλλά και για την ασθενή αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς της πρέπει να στηρίζονται και σε ε, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Πάνω απ' όλα και μιλώ για τις οικογένειες όπου η τραγωδία της ογκολογικής αρρώστιας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σοβαρά στις σχέσεις, σε μια τάση για συγκρούσεις, σε μια τάση για υπερπροστατευτισμό, οδηγεί ως εκ τούτου και σε περισσότερες ε, και, σε, και πέραν των σωματικών προβλημάτων και σε προβλήματα ε, διαπροσωπικά. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ψυχολογική υποστήριξη που θα είναι και αποτελεσματική και που θα προάγει πάνω απ' όλα την ψυχολογική κατάρτιση των, ε, του ιατροφαρμακευτικού ε, προσωπικού. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο οι ψυχολόγοι που θα προσφέρουν αυτή τη βοήθεια, αλλά θα πρέπει σε κάθε στάδιο της παρέμβασης, της παροχής των συμβουλών, ε, στις διάφορες φάσεις της διάγνωσης της αρρώστιας ή της επικοινωνίας, της ενημέρωσης δηλαδή για το αποτέλεσμα της διάγνωσης, πρέπει να υπάρχει αυτή η ψυχολογική υποστήριξη σε όλους τους τομείς των επαγγελματιών της υγείας. Πρέπει και να υπάρχουν ε, κριτήρια για την διάγνωση και για την ε, παραπομπή σε ψυχολογική υποστήριξη για τις ασθενείς, ε, αυτοματοποιημένη κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται η ίδια η ασθενής να αντιληφθεί ότι χρειάζεται την ψυχολογική υποστήριξη και να τη ζητήσει. Στόχος θα πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα ενός προσώπου, μιας ομάδας προσώπων να σταθεί και να, να, σταθεί και να συμπεριφερθεί θετικά απέναντι στα γεγονότα, να μην καμφθεί δηλαδή από μια ε, διάγνωση όγκου, αλλά να ε, αναζητήσει και να βρει τις στρατηγικές που θα είναι πρόσφορες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσα στο πλαίσιο μιας οικογένειας θετικής και ανοιχτής. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very Σας ευχαριστούμε Κύριε Καμπιτέλη. Νομίζω μας ε, επισημάνατε κάποια, από πολύ ουσιαστικά και ε, δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, κυρίως με καρκίνο στο αναπαραγωγικό του σύστημα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γουέντι Γιάρετ, που είναι Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντικαρκυνικών Συλλόγων. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την παρουσίασή μου, μπορείτε να την ε, προχωρήσετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε μια οργάνωση στην οποία συγκεντρώνονται διάφοροι αντικαρκυνικοί σύλλογοι εθνικού επίπεδου. Ε, συμμετέχουν ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Γαλλία, για παράδειγμα είναι η La στην Ιταλία επίσης. Πρόκειται για οργανώσεις δηλαδή που τη σέβεται πολύ ο κόσμος. Και τα έσοδα είναι έσοδα που προέρχονται από εμένα, από εσά, από τους Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή. Αν φαντάζεστε ότι έχουν 15-100 εκατομμύρια, είναι πάρα πολλά χρήματα για να καταφέρει κανείς να συγκεντρώσει και καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος τα δίνει επειδή ακριβώς εμπιστεύεται τους συλλόγους αυτούς. Πώς θα προχωρήσω τις διαφάνειες, ρωτάω μιλήτρια. Οι διάφορες λοιπόν αντικαρκυνικές οργανώσεις ασχολούνται με την πρόληψη, με την έρευνα και τη θεραπεία. Όπως επίσης και την παρηγορητική φροντίδα, όπως έλεγε και η προλαλήσασα, δηλαδή μετά τη διάγνωση ε, βοηθούν τον κόσμο, δίνουν ενημέρωση στο κοινό. Έχουμε να κάνουμε με πολλά είδη καρκίνου και του εντέρου αλλά και πολλά άλλα είδη. Στους χώρους εργασίας επικεντρωνόμαστε επίσης σε κάθε χώρα, φροντίζουμε δηλαδή για την πρόληψη, αλλά συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και με άλλους σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή μιλάμε για τον ε, καρκίνο του στήθους βέβαια, που είναι πολύ συχνός και δυστυχώς η συνάδελφος από το Eurodan δεν είναι εδώ. Αν ήταν εδώ θα μπορούσε να σας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι εγώ για τους καρκίνους που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες πιο συγκεκριμένα. Η δικιά μου οργάνωση λοιπόν, ξεκινήσαμε το 1980, 40 χρόνια σχεδόν τώρα υπάρχουμε. Και δημιουργηθήκαμε ακριβώς επειδή διάφορες επιμέρους ενώσεις αντικαρκυνικές θέλανε να φτιάξουν κάτι μαζί για να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους πιο εύκολα να μην μένει καθεμία στη γωνιά της σε εθνικό επίπεδο. Η γραμματεία μας εδρεύει εδώ, στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εποφελούμαστε δηλαδή από το γεγονό ότι η έδρα μα βρίσκεται εδώ στι Βρυξέλλε. Είμαστε πολύ περήφανοι επίση, γιατί ε, κάποιοι ευρωβουλευτέ που έχουν φτιάξει μια ομάδα που είναι ευρωβουλευτέ κατά του καρκίνου χρησιμοποιούν τη δικιά μα γραμματεία για ενημέρωση και μπορείτε να το βρείτε αυτό MEPs Against Cancer αν ε, το γκουγκλάρετε αυτό θα βρείτε περί τίνος πρόκειται. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν έκλεισαν 10 χρόνια που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ο κύριος Πέτερλε από την Σλοβενία που ήταν πρωθυπουργό της Σλοβενία νωρίτερα είναι πρόεδρος ε, της ε, ομάδας αυτής. Συνεργαζόμαστε λοιπόν μαζί τους αλλά και με άλλους ευρωβουλευτές. Κάθε φορά δηλαδή που ένας ευρωβουλευτές θέλει κάποια ενημέρωση από μας, εμείς φροντίζουμε μέσω της γραμματείας μας να τους εξυπηρετήσουμε. Να λέω next και τότε θα προχωράτε τις διαφάνειες. Καλώς. Λοιπόν, να ο χάρτης που δείχνει πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη, όχι μόνο τον 28, σύντομα 27, αλλά βρισκόμαστε γενικότερα στην Ευρώπη με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα λοιπόν ποιοι είμαστε. Οι οργανώσεις μας έχουν πάνω από 6.000 προσωπικό, πολλούς εθελοντές που χρειάζονται για να βοηθούν. Και αποτελούμε και μια πλατφόρμα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε πολλά να μάθουμε ένα από τον άλλον. Κάτι που συμβαίνει σε μια χώρα μπορεί να βοηθήσει μια άλλη και να μην γίνονται και επικαλύψει. Κάποια στατιστικά δεδομένα τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα νούμερα Πάντως πρέπει να σας πω ότι τα περιστατικά έχουμε στο μεγάλο κύκλο και την θνησιμότητα. Ο καρκίνος του στήθους είναι η πιο σημαντική αριθμή, πιο μεγάλη αριθμή. Ο ορθοκολικός επίσης καρκίνος έρχεται στη δεύτερη περίπτωση. Και μετά έχουμε στα διάφορα έχουμε ε, είτε του σηκωτιού, είτε δέρματος, είτε άλλες περιπτώσεις καρκίνου. Ο καρκίνος είναι υπεύθυνο για 1,3 εκατομμύρια θανάτους το 2010. 26% του συνόλου των θανάτων. Ε, οι άνθρωποι πεθαίνουν πρώτα απ' όλα εξαιτίας καρδιοαγκιακών παθήσεων και η δεύτερη αιτία είναι ο καρκίνος. Έχουμε 760.000 θανάτους για τους άντρες. Για τις ε, γυναίκες τα μεγαλύτερα ποσοστά τα είχαμε στην Ουγγαρία και τη Δανία, όπου εκεί είναι πάνω από 250 θάνατοι για κάθε 100.000 κατοίκους. Τώρα, ποια είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, για τον έλεγχο του καρκίνου. Πριν από 30 χρόνια υπήρχε το πρόγραμμα Ευρώπη κατά του καρκίνου, με ένα πρώτο πρόγραμμα δράσης που έλαβε χώρα το 1987 με το 1989 και ανανεώθηκε με το δεύτερο πρόγραμμα δράσης που πήγε από το 1990 μέχρι το 1994. Βλέπετε εδώ τις δράσεις αυτές για την καταπολέμηση του καρκίνου στις γυναίκες. Τραχύλου, λέμε πώς μπορεί να αποφευθεί, όπως είπε και οι συνάδελφος είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να έχουν ενημέρωση για το πώς μπορούν να αποφύγουν τον καρκίνο. Υπήρχε μια πολύ γνωστή έκθεση για τον καρκίνο του στήθους από Ιταλό συνάδελφο Βερονίτσι. Και χρησιμοποιήθηκε πολύ και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα δράσης κατά του καρκίνου. Τώρα, πρόσφατα, ενώ από το 2011 και μετά, στην πραγματικότητα το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι επιτέλους έφτασε ο καιρός να κάνουμε κάτι παραπάνω κατά του καρκίνου. Τίποτα δεν είχε γίνει από το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε λήξει το 2004, οπότε το 2009 έγινε εδώ στις Βρυξέλλες μια μεγάλη συνάντηση με πολλούς δίψ ε, που όλοι είπαν ότι κάτι πρέπει να γίνει παραπάνω. Οπότε από το 2009 και μετά άρχισαν οι συζητήσεις. Και το αποτέλεσμα ήταν κοινή δράση ε, που ονομάστηκε European Partnership Action κατά του καρκίνου. Ε, πρόκειται για μια δράση πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνήθω ηγούνται οι χώρε μέλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτή τη φορά ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δηλαδή μπόρεσαν να κάνουν κάτι και οι χώρες μέλη και με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτή την κοινή δράση λοιπόν 2011-2014 ο σύνδεσμος αντικαρκινικός πήρε διάφορα μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη του καρκίνου. Το 2011 για παράδειγμα οργανώσαμε σε πολλά μέρη της Ευρώπης κάποιες εκδηλώσεις, flash mobs, και εδώ έχετε τη φωτογραφία, το ονομάσαμε αυτό χορεύοντας για την πρόληψη του καρκίνου. Και καλέσαμε φοιτητέ, νέες γυναίκες να έρθουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε και με το Ινστιτούτο Γυναικών για την Υγεία των Γυναικών που και εδώ είχαμε μία δράση που την ονομάσαμε «Σταματώντας τον καρκίνο πριν να μας σταματήσει αυτός». Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν μέχρι το 2014 και τότε είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις δράσεις για τον έλεγχο του καρκίνου με μια άλλη κοινή δράση, η οποία έλαβε χώρα από το 2014 μέχρι τώρα το 2017. Αυτή η κοινή δράση ονομάστηκε έλεγχος του καρκίνου. το πιο βασικό υπάρχει και στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάτε στο cancercontrol.eu και θα δείτε εκεί ποια είναι τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν στις διάφορες χώρες μέλη. Υπάρχουν πληροφορίες για το τι πρέπει να περιλάβει κανείς ε, σαν ε, πρόγραμμα στη χώρα του. Και το Φεβρουάριο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε αυτή η δράση και εμείς συμμετείχαμε πάρα πολύ σε αυτήν. Υπήρξαν διάφορα έγγραφα πολιτικής το οποίο εκπονήθηκαν στα πλαίσια αυτή τη δράση και καταλήξαμε και σε συστάσει για την αντιμετώπιση του καρκίνου στη γυναίκα. Αυτέ εδώ που βλέπετε είναι οι συστάσει για τι γυναίκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μην ξεκινάτε συνολική ακτινολογική θεραπεία για το στήθος σε μια κλασματοπία 25 σαν μέρος θεραπείας ή συντήρησης εφόσον η γυναίκα είναι πάνω από τα 50 και βρίσκεται σε ένα αρχικό στάδιο επιθετικού καρκίνου του στήθους να βοηθήσουμε επίσης να γίνεται έλεγχος για τον καρκίνο και σε μετανάστριες. Επίσης να υπάρχει ενημέρωση με κινητά επιτελεία ώστε να μπορούν οι γυναίκες παντού όσο απόκεντρα και αν ζουν να ελεγχθούν για τον καρκίνο. Και το άλλο ήταν να στηρίξουμε πολιτικές που βοηθούν τις γυναίκες οι οποίες φροντίζουν ασθενείς, καρκινοπαθείς, τι να κάνουν και πώς να τους φροντίσουν ακριβώς. Γιατί καλά φροντίζεις εσύ και αν και εσύ όμως Τι κάνεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στήριξη και για τους ανθρώπους αυτούς που φροντίζουν άλλους. Ε, μητέρες, για οτιδήποτε. Πολύ δουλειά είχαμε να κάνουμε. Μια άλλη κοινή δράση επίσης ξεκίνησε στη συνέχεια. Τώρα εδώ θέλω να δούμε λιγάκι τον Ευρωπαϊκό Κώδικα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ξεκίνησε ήδη από το 1987 και προχώρησε σιγά σιγά φυσικά με διάφορες ενημερώσεις, αναθεωρήσεις κτλ. Είναι κάποια μηνύματα που στόχο έχουν το κοινό προκειμένου να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν τον ε, καρκίνο. Βασίζονται σε στοιχεία από την ε, Διεθνή Οργάνωση Υγείας και χρηματοδοτήθηκε η εκστρατεία αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ο κώδικας αυτός επικεντρώνεται σε δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι πολίτες για να αποφύγουν τον καρκίνο. Κάποιες μικρές προτασούλες είναι δηλαδή πολύ φιλικά διατυπωμένες για να μπορεί και ο κόσμος να πάρει το μήνυμα εύκολα. Λέει ας πούμε μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε καθόλου προϊόντα καπνού. Ε, φροντίστε στο σπίτι σας να μην ε, καπνίζετε. Στηρίξτε όλες τις πολιτικές που είναι ε, αντικαπνιστικές και στους χώρους εργασίας σας. Εδώ, στο Κοινοβούλιο για παράδειγμα, που έχει γίνει. Έπειτα λέμε τρώτε υγιεινά, ε, τρώτε πολύ σπορά προϊόντα, ε, περιορίστε στη διατροφή σας ε, υψηλής θερμιδικής αξίας προϊόντα, αλκοόλ, μην πίνετε αλκοόλ και αν πίνετε ελαχιστοποιήστε το. Είναι καλύτερα για να αποφύγετε τον καρκίνο να μην πίνετε καθόλου αλκοόλ. Αποφύγετε τον ήλιο, κυρίως για τα παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε σολάριο και στο χώρο εργασίας να προστατεύετε τον εαυτό σας και αν ε, και φροντίστε να μην ε, υποβάλλεστε σε ακτινοβολία. Αυτά γενικώ. Και μετά συγκεκριμένα για τις γυναίκες λέμε ότι ο θυλασμός μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Οπότε αν μπορείτε θυλάστε το παιδί σας. Έπειτα, οι ορμονικέ ε, θεραπείες υποκατάστατου στην ε, κλιμακτήριο αυξάνουν τον κίνδυνο για κάποιους ε, καρκίνους. Οπότε αποφύγετε τέτοιε θεραπείε. Φροντίστε τα παιδιά σα να εμβολιάζονται για την υπατήτηδα Β, για το ανθρώπινο θύλωμα επίσης. Επίσης συμμετέχετε σε προγράμματα ε, για τη διάγνωση του καρκίνου. Είτε πρόκειται για το έντονο, είτε πρόκειται για το στήθος, είτε για το ορθοκολικό καρκίνο. Τώρα θέλω να έρθω λίγο πίσω όσον αφορά την οδηγία που δώσαμε για τα σολάριου. Κυρίως οι γυναίκες νέες ή μεσήλικες χρησιμοποιούν ε, τα σολάριου. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλάει για την εκτινοβολία αυτή και αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα τα σολάριου, τα οποία χρησιμοποιούνται όχι βέβαια για λόγου υγείας, όταν χρησιμοποιούνται επειδή θέλει μια γυναίκα να φαίνεται πιο μαυρισμένη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το συμπέρασμα της έκθεσης αυτής είναι ότι οποιοδήποτε είδους τέτοια περίοδος εκτινοβολία και αυτή η, την οποία λαμβάνουμε στα σολάριου είναι ιδιαίτερα βλαβερή γιατί και προκαλεί καρκίνο και τον ε, επιδεινώνει. Μελανόματα παρουσιάζονται. Κυταρικό καρκίνωμα. Ακούμε τέτοια επιχειρήματα πολλές φορές από τα σολάριου που λένε ότι όχι, είναι καλά γιατί χρειαζόμαστε τις βιταμίνες που μας δίνουν. Όχι όμως. Εμείς έχουμε αποδείξεις, επιστημονικά δεδομένα που λένε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή ότι τα υπέρ δεν είναι όπως τα διαφημίζουν οι σχετικές επιχειρήσεις. Και στο κάτω-κάτω, άμα θέλετε βιταμίνη Δ, D, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να την απορροφήσετε. Δεν χρειάζεται να πάτε στα σολάριουμ και να πάτε να εκτεθείτε σε περίοδες ακτινοβολίας. Είναι σαν να έχετε έγκαυμα τάξης του 12. Όταν ακούμε ότι έχουμε πολύ ήλιο και ότι τα επίπεδα είναι στο 12, ε, μας το λένε για να προστατευτούμε, γιατί σημαίνει ότι είναι ανισχυτικό. Ε, λοιπόν, στα σολάρια πάντα έτσι είναι. Άλλες δράσεις τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα κοινό ερευνητικό κέντρο που είναι εκείνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μιλάνο, όπου έχουν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του καρκίνου του στήθους. Είναι μια δράση που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια. Ε, συνάδελφος βέβαια θα σας πει περισσότερα για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του καρκίνου. Αυτό όμως που θέλω να σας πω εγώ είναι να σας μιλήσω για μια άλλη νέα κοινή δράση για τον εμβολιασμό που αρχίζει του χρόνου. Δεν είναι ειδικά για τον καρκίνο, είναι εκστρατεία εμβολιασμού για διάφορα πράγματα. Συνεργαζόμαστε με το Γαλλικό Υπουργείο πάνω σε αυτό και θα επικεντρωθούμε σε δύο από τα μηνύματα που σας ανέφερα μέχρι τώρα που έχει να κάνει εμβολιασμό για, κατά της υπατήτηδας Β και κατά του ανθρώπινου θυλώματος. Πολύ σύντομα λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά σε πολλές χώρες όσον αφορά τον εμβολιασμό έχουν πέσει τα επίπεδα. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα στα μέσα ενημέρωσης, διαδόσεις, ότι ο εμβολιασμός οδηγεί σε αυτισμό ή δεν ξέρω εγώ σε τι άλλα προβλήματα. Και τα μέσα ενημέρωσης αυτό το πήραν, το κυκλοφόρησαν πολύ και είναι κάποιοι γονείς που δεν θέλουν να εμβολιάζουν τα παιδιά τους κατά της επατήτηδας Β. Και Γι' αυτό τώρα εμείς έχουμε αυτή την κοινή δράση για τον εμβολιασμό. Αναφέρθηκα στην ομάδα Ευρωβουλευτών κατά του καρκίνου. Έχουν ιστοσελίδα και θα δείτε ποιοι είναι οι στόχοι τους εκεί. Εμείς συνεργαζόμαστε με όσο μπορούμε περισσότερους ευρωβουλευτές Έρχονται καμιά φορά ευρωβουλευτέ μα, ρωτάνε κάτι για τον έλεγχο ε, του καρκίνου και εμεί του βοηθούμε με στοιχεία, με συμβουλέ πώ να διατυπώσουν ε, την ε, θέση τους, την τοποθέτησή τους. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μου είπαν ότι πρέπει να περάσουμε κατευθείαν στην Current Μπεντ. Είναι αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της οργάνωση Europa Donna μια αντικαρκυνικής οργάνωση που ασχολείται ιδιαίτερα με τον καρκίνο του μαστού. Η έδρα τους βρίσκεται στο Μιλάνο, αλλά έχουν παραρτήματα σε όλη την Ευρώπη. Η, ομάδα, η οργάνωση Europa παρτίζεται απαρτίζεται από 47 χώρε μέλη, στην οποία συμμετέχουν όλε οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε εδώ τον κατάλογο με τι 47 χώρε που συμμετέχουν στην οργάνωση Europa Και μέσα στα 22 χρόνια άλλαξε η αποστολή, δηλαδή σκοπό του είναι να φροντίσουν πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων σε σωστή ενημέρωση, ποιοτικό προληπτικό έλεγχο, διάγνωση και θεραπευτική αγωγή. Δηλαδή καλύπτουν όλε τι πτυχέ του καρκίνου του μαστού. Μερικά στοιχεία που αφορούν τον καρκίνο του μαστού τα, η συχνότητα. Αναφέρθηκα πολλέ φορές τα ποσοστά. Είναι ο πιο κοινό καρκίνο ο καρκίνο του μαστού στις Ευρωπαίε. Μάλιστα το 2012 ήταν 494.000 395.000 τα περιστατικά, ενώ στην Ευρώπη των 28, 361.600 τα περιστατικά καρκίνο του μαστού. Μία στις 8 γυναίκες στι 28 χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωση θα εμφανίσουν καρκίνο πριν το 85. 20% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού στην Ευρώπη εμφανίζονται σε γυναίκες κάτω των 50 και 37% σε γυναίκες μεταξύ 50 και 64 ετών. Οι υπόλοιποι καρκίνοι του μαστού εμφανίζονται μετά τα 64. Σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα και την επιβίωση, ο καρκίνο του μαστού έχει την υψηλότερη θνησιμότητα κάθε άλλη μορφή καρκίνου παγκοσμίω αλλά και στην Ευρώπη. Ο, ο αριθμό των γυναικών που υπολογίζονται ότι έχουν χάσει τη ζωή του από τον καρκίνο του μαστού το 2012 στην Ευρώπη ήταν 143.000 περίπου και στι 28 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση 91.000. Και μάλιστα η σχετική επιβίωση πενταετής ε, γυναικών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού είναι 80%. Δηλαδή το 80% των γυναικών που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού ε, παραμένουν ζωντανές μετά από μία πενταετία από τη διάγνωση, που σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί καλή θεραπεία μετά τη διάγνωση και να επιβιώσουν και μετά τη θεραπεία. Τι επιζητεί η οργάνωση Europa Donna. Θέλουν να, εξασφαλίσουν την, τον καλύτερο προληπτικό έλεγχο και θεραπεία για τις γυναίκες και μάλιστα θέλουν ε, σωστές, ακριβείς και ενημερωμένες ε, πληροφορίες. Θέλουν την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή και πρόσβαση των γυναικών στις σχετικές ακριβείς πληροφορίες και επίσης ε, να προσφέρονται όλες αυτές οι υπηρεσίες από τα εθνικά συστήματα υγείας ποια είναι τα προσκόμματα σε μια βέλτιστη παροχή υπηρεσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικά επίπεδα στα κράτη-μέλη, διαφορετικά συστήματα υγείας των κρατών μελών. Υπάρχουν τεράστιες διακοιμάσεις και διαφορές, οπότε η πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή και στα, στα συστήματα υγείας διαφέρει πολύ αισθητά μερικές φορές, ακόμη και στις περιφέρειες ενός κράτους μέλους. Και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και προδιαγραφές δεν είναι κοινά τα, οι απαιτήσει για τα ειδικευμένα ιδρύματα, τα δικαρκυνικά. Επίσης, ε, κλειστό το ιατρικό κατεστημένο και πώς μπορούμε να διευρύνουμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Η πολιτική της Παντώνα είναι να εξασφαλίσει υπηρεσίες ε, χάρη των καρκινοπαθών, ώστε ε, να φτάσουμε σε ποιοτικέ προδιαγραφέ χάρη στην ανάπτυξη πολιτικών. Έχουμε λοιπόν παραρτήματα τη οργάνωση Γερό Παντώνα σε όλε τι χώρε που παρέχουν σημαντικέ πληροφορίε και συνεργάζονται προκειμένου να επηρεάσουν του πολιτικού την ομοθεσία, τους κανονισμού, ακόμη και την οτροπία μέσω του λόμπι που κάνουν ε, για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Συνεργάζονται με πολλούς συμφεροντούχους και ενδιαφερόμενους. Βλέπετε ότι είναι πολύ δραστήρια η οργάνωση αυτή δεν πρόκειται να σας διαβάσω όλα αυτά τα ακρονίμια. Η IRC είναι ε, από το Ερευνητικό Κέντρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Έχουμε μια ε, οργάνωση νοσηλευτών, έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, οργανώσεις που έχουν παρατήματα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οργανώνουν την παγκόσμια, την ημέρα της, ε, του καρκίνου του μαστού, η εκδήλωση που έγινε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, σε σχέση με τη συνεργασία τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2001 και 2002 είχαν ε, συναντήσει με εμπειρογνώμονες. Το 2003 βοήθησαν ε, για τη, στη διαμόρφωση του, της σύστασης του Συμβουλίου για τον προληπτικό έλεγχο. Επίσης βοήθησαν να εκπονηθεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καρκίνο του μαστού και το 2006 συμμετείχαν στο δεύτερο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καρκίνο του μαστού και μάλιστα την ίδια χρονιά είχαν την τέταρτη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2010 είχαν τη δράση Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του καρκίνου του μαστού και ένα ε, σύστημα ευρωπαϊκής πιστοποίησης για τα SBUs που δεν ξέρω τι σημαίνουν. Επίσης, έχουμε το Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, πρωτοβουλία που έλαβε για τον καρκίνο του μαστού. Ξεκίνησαν ε, σχετικές ε, διαπραγματεύσεις και μάλιστα είχαμε και την σχετική γραπτή δήλωση το 2015 από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και το 2017 έχουμε τις εκθέσεις για την εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου. Τώρα, ποιε είναι οι βασικέ προτεραιότητε που εδράζονται πια στην πολιτική. Εφαρμογή είναι το σημαντικό. Ε, Προληπτικό έλεγχο με βάση τη μαστογραφία, κατευθυντήριε γραμμέ και ψηφίσματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2003 μέχρι το 2006, ειδικέ μονάδε για τον καρκίνο του μαστού, η ευρωπαϊκή πιστοποίηση και ε, βεβαίως ποιότητα του συστήματο για τι υπηρεσίε καρκίνου του μαστού. Αυτά απορρέουν όλοι από την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τον καρκίνο του μαστού. Εδώ έχουμε τι ε, ε του γράφου για το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά του καρκίνο του μαστού. Βλέπετε τι ευρωβουλευτέ και του ευρωβουλευτέ που υπέγραψαν αυτή την κοινή διακήρυξη. Το 2010 και 2015 έγινε γραπτή διακήρυξη για τον καρκίνο του μαστού, ώστε να παραμείνει σημαντική προτεραιότητα το πρόγραμμα Υγεία Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε την δήλωση για τον προληπτικό έλεγχο μέσω τη μαστογραφία και την ανάγκη να, υπάρχει δική μονάδα για τον καρκίνο του μαστού. Ε, εφαρμογή από το 2016 και έχουμε κάποιε πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών και την πιστοποίηση των ε, μονάδων μαστού μεταστατικός καρκίνος του μαστού και ε, ψυχολογική ε, αρρωγή που είναι πολύ σημαντική όπως ακούσαμε. Αυτή είναι η τέταρτη δημοσίευση των καθεδιογραμμών του 2006 που ε, περιγράφουν τις καλύτερες πρακτικές, θεσπίζουν πρότυπα που ζητούν να είναι αμερόληπτα και μετρήσιμα. Οπότε ασχολούνται με πολιτική, εκστρατείε, ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση στι γυναίκε. Και αυτό είναι ένα σύντομο οδηγό των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Γραμμών. Αν δείτε τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο... το σχετικό έγγραφο είναι πολυσέλιδο. Γι' αυτό και η Europa Donna και με εντυπωσίασε με την προσπάθεια κλαίκευση που κάνει, συνέταξε ένα πολύ σύντομο, μια σύνοψη αυτού του οδηγού, μια επιτομή, αν θέλετε, αυτού του οδηγού των κατευθυντηρίων γραμμών, που είναι πολύ πιο προσιτό στο κοινό. Επανέρχομαι τώρα στην, στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το καρκίνο του μαστού, που αναπτύχθηκε εξαιτία σημαντικών και συνεχών ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τη συχνότητα, τη θνησιμότητα, τον επιπολασμό και την επιβίωση από καρκίνο του μαστίου σε πολλές χώρες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιωθεί και να αρμονιστεί η περίθαλψη για κρούσματα περιπτώσει καρκίνου του μαστού στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας ε, σημαντική, σημαντικό ποιοτικό σύστημα για υπηρεσίες ε, καρκίνου του μαστού με σωστή πιστοποίηση, υψηλή ποιότητα, ε, σημαντικές αποδείξεις επιστημονικά και απορίσματα και ενημέρωση συνεχή των καθεδρίο γραμμών. Και μάλιστα γίνεται συντονισμό ε, τη πρωτοβουλία αυτή από το Κοινό Κέντρο Ερευνών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεται λίγο έξω από το Μιλάνο. Συμμετέχουν 70 ε, εμπειρογνώμονε με επαγγελματίε καρκινοπαθεί σε δύο ομάδε εργασία. Έχουμε την ε, ομάδα ανάπτυξη των καθεφιδίων γραμμών και την ομάδα ανάπτυξη του συστήματο ε, βεβαίω ποιότητα. Και έχουμε 35 χώρε ε, της 28 ης Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ισλανδία, ε, η Ισλανδία το Φι, τη Φιρόμ, το Παυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία. Ε, Υψηλότερε είναι οι προσδοκίε γιατί στόχο τη πρωτοβουλία είναι να έχουμε νέε κατευθυντήριε γραμμέ Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επικαιροποιούνται συνεχώ, θα βρίσκονται φυσικά πρόσθετε στο διαδίκτυο και είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο αυτό το έργο, γιατί είναι πολύ συμφεροντούχοι και οι ε, ενδιαφερόμενοι. Πάντως ε, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και την παρακολούθηση και σίγουρα θα πρέπει να είναι σαφείς αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές από τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από τέτοια συστήματα. Θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα, αυτός είναι κοινό στόχος όλων που ενεργοποιούμαστε σε αυτό το τομέα και επίσης ε, υπάρχει ένα ερωτηματικό στο κατά πόσο θα ολοκληρωθούν όλα αυτά μέχρι το 2019, γιατί είναι η συνεργασία με τόσους πολλούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν θα είναι και τόσο εύκολο να ολοκληρωθεί. Και επίσης θέλουμε πανευρωπαϊκή εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Οπότε, ποια είναι η ισχύ της οργάνωσης ε, Europandona. Έχω σαφείς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι μια οργάνωση με εκτεταμένο δίκτυο ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά χρειάζεται ένας κατάλληλος συντονισμός. Και ακόμη και αν επιτύχουμε καλό συντονισμό, θα είναι ε, ε, σημαντικός ο αντίκτυπος στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά συστήματα υγείας. Η Europa Donna θέλει να συνεχίσει ανανέωση αυτή της δέσμευση, αξιοποίηση αυτή της όθηση που έχει δημιουργηθεί στη συνεργασία με τους αντικαρκυνικούς συλλόγους και εταιρείε, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εθνικούς ε, φορείς. Συνεχίζουμε τις ε, συνεργασία μας με την Παντώνα για θέματα καρκίνου του μαστού και πραγματικά εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το έργο αυτής της οργάνωσης γιατί και σε εθνικό επίπεδο οργανώσαμε τις, ε, ομάδες, τις εβδομάδες ευαισθητοποίησης ε, για τον καρκίνο του μαστού και μάλιστα και η Κάρεν ε, είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει απορίε. Μπορώ να τη τηλεφωνήσω και αμέσως σας μεταφέρω τις απαντήσεις της. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε περίπου 15 λεπτά στη θέση μας για ερωτήσεις και σχόλια. Αν έχετε κάτι για τις ομιλήτριες, την Κάρεν Μπέν. Εδώ η ευκαιρία. Θέλει κανείς καμία να λάβει το λόγο. Κυρία Ward. Ζητώντας συγγνώμη που έφτασα τόσο αργά. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί με απασχολεί και στην οικογένειά μου και η αδελφή μου έχει επιβιώσει από καρκινό του μαστού. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν αυτή η μελέτη που δεν πρόλαβα να παρακολουθούσω μιλούσε και για πρόληψη, πιθανά αίτια ή μιλούσε μόνο για διάγνωση. γιατί είναι τόσοι οι άγνωστοι παράγοντες. Που θα πρέπει να είναι πιο γνωστοί για να μπορούμε να του αντιμετωπίσουμε. Επομένω είναι κάτι που αφορά και τη διάγνωση και το περιορισμό ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τον προληπτικό έλεγχο, άλλους παράγοντες. Κυρία Γιάρετ, εννοείται το κέντρο έρευνας. Ναι, έφτασα, έφτασα με καθυστέρηση και ίσως κάτι δεν κατάλαβα καλά και στο συγγνώμη. Ή αν μου ξέφυγε κάτι. Αλλά το κομμάτι που παρακολούθησα μου έδωσε την εντύπωση ότι αναφερόταν κυρίως στην αναγνώριση του προληπτικού ελέγχου και των αγωγών. Αλλά θα ήθελα να κοιτάξουμε και τους ε, και τα αίτια, του επιβαρυντικού παράγοντε και να ρωτήσω βέβαια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα Ευρώπη κατά του καρκίνου που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια έχει κοινέ δράσεις αναπτύξει με δότη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, φτάσαμε στην ε, επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του καρκίνου, του ΣΥΑΡΚ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και συγκεκριμένα, αν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα στη διαφάνεια, στο σημείο που αφορά την πρόληψη, γιατί κάνατε λόγο και για ε, υποστήριξη, υπηρεσία υποστήριξης. Οι συνάδελφο μίλησαν νωρίτερα για το θέμα αυτό. Χάσατε τη δική τη την παρουσίαση. Πάντω για μα της Ευρωπαϊκής Ενώσης κατά του καρκίνου. Έχουμε ομάδα εργασία για την υποστήριξη των ασθενών με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση αυτή, διότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην θεραπεία και την έρευνα. Έχουμε πιο πολλές γυναίκες που έχουν επιβιώσει ε, και χρειάζονται την υποστήριξη αυτή για το τι γίνεται μετά την ε, διάγνωση. Και από τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει, παραδείγματι, είναι αυτά που έχουν να κάνουν και με την ε, με το πώς βλέπει η γυναίκα τον εαυτό της, πώς διαχειρίζεται την, ε, τον οικογενειακό της, τον, ε, τη σχέση της με τον σύντροφό της. Έχουμε σε εθνικό επίπεδο ε, τις ενώσεις για την καταπολέμηση του καρκίνου που εξασφαλίζουν τέτοιου είδους υποστήριξη. Εμείς λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, η ECO, προσφέρουμε διαθέτουμε τις πληροφορίες, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα ε, υποστήριξης και στις προηγούμενες κοινέ δράσεις και στην τωρινή κοινή δράση. Εδώ ακριβώς αναφερόμουν στις συστάσεις που αφορούν τις γυναίκες. Στον ε, οδηγό αυτό συνιστούμε να υπάρχουν ειδικά προγράμματα πλοήγησης για τις γυναίκες και για, την, ε, για τον προληπτικό έλεγχο, αλλά και για την υποστήριξη ε, της ίδιας της γυναίκας ε, των μελών της οικογένειας, όποιον φροντίζουν τις γυναίκες. Πρέπει όμως και εμείς, εμείς οι ενώσεις, να προσέχουμε περισσότερο για να προσφέρουμε αυτήν την υποστήριξη στις ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις ε, ομιλίες σας, για τις παρεμβάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι, εδώ είμαι. Ήθελα μου τρέξει την προσοχή του η αναφορά σε μια εκστρατεία που θέλετε να αναπτύξετε για τα... τις επιφυλάξεις με τους εμβολιασμούς γιατί σε πολλά κράτη γινόμαστε μάρτυρες μιας ε, εκστρατείας ε, κατά των εμβολιασμών. Έχετε δει, εσείς λοιπόν κάτι συγκεκριμένο, έχετε δει κάποιες γυναίκες σε παραδείγματι να αποφεύγουν τη μαστογραφία, γιατί στη Σλοβακία, την πατρίδα μου, υπάρχουν τέτοιου είδους Να μην κάνουν οι γυναίκες μαστογραφία, να μην συμμετέχουν στους προληπτικούς, να μην πηγαίνουν για προληπτικό έλεγχο. Και όταν θέλησα εγώ να καταπολεμήσω αυτή την ε, εκστρατεία, ε, κατηγορήθηκα ότι θέλω να προξενήσω εμφάνιση καρκίνων στις γυναίκες, επειδή υποστηρίζω τη μαστογραφία. Ενώ σώζω τις ζωές με την, προ... με την διάγνωση, με την πρώιμη διάγνωση. Είπατε ότι θα κάνετε λοιπόν μια εκστρατεία ενημέρωσης ε, για του εμβολιασμού για τις μαστογραφίες υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Κύριε Γιάρετ, την κατάσταση στη Σλοβακία δεν την γνωρίζω ε, προσωπικώς. Έχουμε βέβαια ένωση κατά του καρκίνου εκεί. Πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε διμερώς για το πώς μπορεί να ε, δραστηριοποιηθεί και η Σλοβακική μας Ένωση για το θέμα που σας ενδιαφέρει συγκεκριμένα για το αν ε, αυτή τη διστακτικότητα εναντί των προληπτικών ελέγχων που αφορά και τη μαστογραφία ε, σκοπεύουμε να την ε, αντιμετωπίσουμε. Όταν μίλησα για αυτή τη διστακτικότητα αναφέρομαι ιδιαίτερος στη προγράμματα εμβολιασμών. Επομένως δεν αφορά ευθέως τη μαστογραφία. Αλλά με αυτό που μου λέτε και τις ανησυχίες που εκφράσατε για τη Σλοβακία ασφαλώς ε, θα κοιτάξουμε με την ένωσή μας της Σλοβακίας να διερευνήσουμε την κατάσταση, να ενημερωθούμε. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, έχετε κάποια ιδέα. Ε, η έκθεση στην ακτινοβολία. Η απάντηση χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα, έκθεση στην ε, ακτινοβολία. Ναι, κοιτάξτε. Έχουμε πολλούς που έρχονται με τέτοιου είδους ερωτηματικά. Μας λένε, μα είναι ασφαλής η μαστογραφία» εκτιθέμεθα στην ακτινοβολία κτλ. Και η απάντηση που δίνουμε είναι μιλήστε με τον ογκολόγο, με τον γιατρό σας και σταθμίστε τους παράγοντες, γιατί αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, η, η ηλικία που με βάση τις συστάσεις υποδεικνύει την διεξαγωγή, την υποβολή σε μια μαστογραφία, Αλλά πάλι από αυτό που λέτε, οι γυναίκε εκείνε οι οποίε θα έπρεπε με βάση τη στάση να κάνουν μαστογραφία είναι αυτέ που διστάζουν. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι η κατάσταση στη χώρα, γιατί μπορεί και τα ε, μέσα μαζική ενημέρωση να διωγγώνουν ε, τα προβλήματα. Πολύ ευχαριστώ να το συζητήσουμε διμερώ. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρο, δεν βλέπω να ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Η κυρία Καμπιτέλη, παρακαλώ, αν έχει κάτι για να ολοκληρώσει. Σαφές είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια πλήρης ε, υποστήριξη σε ολόκληρη τη διαδικασία της θεραπείας από τη διάγνωση, τις δυνατότητες για θεραπεία, τις δυνατότητες για παρέμβαση, για επέμβαση και πάντως και για αυτή σας την ε, τοποθέτηση για την επιφυλακτικότητα σε σχέση με τη διεξαγωγή μιας διαγνωστικής, με την υποβολή σε μια διαγνωστική μέθοδο όπως ε, η μαστογραφία. Θα μπορούσα από ψυχολογικής έποψης να πω ότι ίσως θα ήταν και ένας λόγος ε, της άρνησης, της έκθεσης των κίνδυνων να διαγνωστεί αυτή η αρρώστια. Ε, γενικά και στη γενετική διάγνωση για τον κίνδυνο της ογκογέννησης. Βλέπουμε μερικές φορές να αλλάζει συμπεριφορά ε, η ομάδα κινδύνου. Φαίνεται δηλαδή να φοβάται να, και ως εκ τούτου να αποφεύγει την ε, υπαγωγή σε αυτή την, την ε, εξέταση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η πλαισίωση στη στο διαγνωστικό τμήμα με την υποστήριξη την ψυχολογική που θα ενημερώσει και για τα ωφέλη και την, τον αντίκτυπο μιας έγκαιρης διάγνωσης. Κυρία Ιούτο, πολύ σύντομα και εγώ θέλω να συμπληρώσω για να ολοκληρώσω. Ε, ήρθαν πολλές συνάδελφοι αφού είχα ήδη διατυπώσει τις ε, προτάσεις μου για την ε, ουσία της έκθεσης, όπως σκοπεύω να διατυπώσω. Και από την αρχή βέβαια της ε, ακρόασης, ή πριν να ξεκινήσει μάλλον η ακρόαση, άκουσα ερωτήσεις σχέση με διάφορες τυπολογίες θεραπείας. Λοιπόν, για να το πω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει μακριά από μένα κάποια σκέψη για διατύπωση έκθεσης που θα κάνει προτάσεις για θεραπείες ογκολογικές. Μακριά από μένα έκθεση, η ιδέα ότι θα διατυπώσω μία έκθεση η οποία θα τοποθετείται υπέρ κατά των εμβολιασμών. Άλλα είναι αυτά τα ζητήματα, ξένα προς εμένα και θα συστηθούν σε άλλους χώρους. Αλλά ας μην χάσουμε την ουσία, ας μην χάσουμε το στόχο που θα έχει αυτή η έκθεση, που είναι να συνοδεύσουμε τη γυναίκα σε όλες αυτές τις πτυχές και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει από τη στιγμή που ασθενεί. Σε πρώτη φάση την υπαγωγή μετά στις θεραπείες και τη φάση που ακολουθεί τις θεραπείες. Δηλαδή αντιμετώπιση σε ευρύτατο φάσμα, σε πλήρες φάσμα της αρρώστιας την επιλογή της ε, ασθενούς ως προς την ε, ε, μονάδα, την ιατροφαρμακευτική, η οποία θα της προσφέρει τις θεραπείες και τις αγωγές. Θέλουμε δηλαδή κάθε γυναίκα να έχει και πρώιμη πρόσβαση, αλλά πάνω απ' όλα και ψυχολογική υποστήριξη, εκεί όπου είδαμε υπάρχουν πολύ μεγάλα ευτυχώς ποσοστά επιβίωσης, Ευτυχώ μεν, που όμω ταυτόχρονα απαιτούν και σημαντική ψυχολογική υποστήριξη. Δεν είναι δεύτερη σημασία σε αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Είναι εκ των όνων κάνευ και αυτό ακριβώ θέλω να τονίσω και ε, ελπίζω κατά την επεξεργασία της, ε, της έκθεσης και των τροπολογιών ε, να μην λησμονήσουμε αυτόν τον στόχο γιατί βεβαίως είμαστε η κατ' ουσίαν επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα αυτά μεν, αλλά α μην συζητήσουμε θέματα τα οποία δεν αλήκουν στην θεματολογία αυτής τη έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εσείς θέλετε να καταλήξετε σε συμπεράσματα, Παρατηρήσει. Νομίζω ότι είπα αρκετά, λέει η κυρία Γιάρετ, αλλά σίγουρα δεν έχουμε κάνει αρκετά στον τομέα της πρόληψης. Είπε η πρόεδρος ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές, την πρόσβαση, στην ε, φροντίδα και θα έλεγα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο το θέμα της πρόληψης του καρκίνου. Τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ακολουθώντας τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του καρκίνου. Ξέρω, είπατε ότι στην έκθεσή σας δεν θα αναφέρετε θεραπείες, ναι. Μιλάμε όμως για την ισότητα στην πρόσβαση. Πρόσβαση σε φάρμακα, όταν κάποιος διαγνωστεί καρκινοπαθής, θέλει να θεραπευτεί αμέσως, να έχει πρόσβαση στη θεραπεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί όμως. Μπορεί να υπάρχει μια θεραπεία διαθέσιμη σε μια γειτονική χώρα και κάποιος άλλος ασθενής σε άλλη χώρα να μην έχει πρόσβαση σε αυτήν. Οπότε πρέπει να δούμε όλο το φάσμα θα κοιτάξουμε φυσικά την έκθεσή σας. Καλό θα ήταν αν μπορούσατε να πείτε κάτι και για αυτό το θέμα της πρόσβασης στη θεραπεία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία, έτσι εδώ ολοκληρώνεται η ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν. δεν Κάραν δεν μπόρεσε να έρθει εδώ, αλλά η συμβολή της έγινε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και θα επανέλθουμε δίχως άλλο θα συζητήσουμε την έκθεση όταν θα έχουμε τροπολογίες, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι προσωρινό. Είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Ε, πρέπει όντως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πρόληψη κατά του καρκίνου. Φοβάμαι ότι θα χρειαστεί πολλή χρόνο ακόμα μέχρι να μπορούμε να πούμε ότι τον νικήσαμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε λοιπόν εδώ σε αυτή την ακρόαση. Μπορείτε να παραμείνετε αλλά απ' την άλλη ε, πρέπει να φύγετε. Εμείς θα συνεχίσουμε με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Συνεχίζουμε με τις εργασίες μας και πριν περάσουμε στις εκθέσεις θα θέλω να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεών μας στις 12 Ιουλίου και τις 4 Σεπτεμβρίου. Συμφωνείτε? Ωραία. Και τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση, είναι το σημείο 5 στην εμμυρίσια διάταξη. Πρόκειται για γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη. Η συγκήτριά μας είναι η Λίνεα Έγκστρομ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα μιλήσω σου ειδικά, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό, γιατί έχουμε στη Βόνη το Νοέμβριο την επόμενη διάσκεψη για το κλίμα. Αρχίζω λοιπόν με το υπόβαθρο και γιατί ανέλαβα αυτή την έκθεση. Και θέλω επίσης να πω ότι διακόπτει η Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη γαλλική διερμηνία φαίνεται. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα είναι εντάξει, συγγνώμη. Ωραία. Ε, συνεχίζω λοιπόν είναι, λέγαμε, πρόβλημα το θέμα αυτό της κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι ακόμα πιο μεγάλο για αυτούς που δεν έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ε, φυσικές καταστροφές κλπ. Πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε πολύ, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για την ευθύνη που θα δείξουμε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαιώματο στην υγεία, πώς οι τοπικές κοινότητες θα έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία να συνεχίσουν να υπάρχουν. Φυσικά και χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες και περισσότερη ισότητα μεταξύ διαφορετικών γενεών. Η κλιματική αλλαγή και ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους. Να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία, να υποφεληθούμε από τα ωφέλη. Στην ε, υποσαχάρια Αφρική, την Ασία, πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν εξαιτίας ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Η σύμβαση του ΟΗΕ για να αποφευθεί η απερίμωση λέει ότι 25 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν στο μέλλον να εγκαταλείψουν τη γη τους και το 2050 θα είναι 200 εκατομμύρια άνθρωποι που θα ονομάζονται πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό και μιλάμε για την κλιματική δικαιοσύνη. Και οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο. Είναι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες αναγκάζονται περισσότερο να εγκαταλείψουν την γη τους, τα μέρη τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αυτή λοιπόν θα αναγκάσει τον κόσμο όλο και περισσότερο να φεύγει από τα σπίτια του. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση στο μέλλον και χρειάζεται μια συνολική σφαιρική στρατηγική για να αντιμετωπιστεί. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕΠ, έχει περάσει μηνύματα για την κλιματική αλλαγή η ατζέντα του 2030 και η Συμφωνία των Παρισίων αποτελούν νομικά πλαίσια προκειμένου να εκπονηθεί παρετέρω νομοθεσία και να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ένα νομικό πλαίσιο που λέει ότι πρέπει να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις πολιτικές μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Άρα και εδώ πρέπει να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες απέναντι σε αυτή την κλιματική αλλαγή για όλους. Πρέπει να στηρίξουμε την κλιματική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη και να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες αυτούς που έγιναν πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια. Πάντα στα πλαίσια του ΟΗΕ και της διάσκευσης για το κλίμα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Γιατί δηλαδή ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή. Τώρα όμως έρχομαι στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ε, για τις οποίες μιλάμε στην έκθεσή μου. Και λέω πρώτα απ' όλα ότι οποιοδήποτε έχει συνυπογράψει τη Συμφωνία των Παρισίων το έκαναν σε θελοντική βάση. Όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ισότητα, η ισότητα απέναντι στις κλιματική αλλαγή, ας πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Στις συνθήκες αναφέρεται ως στόχος αυτή η ισότητα. Οπότε αυτήν πρέπει να την προάγουμε. Και θέλω να τονίσω και κάτι για την επόμενη διάσκεψη για το κλίμα που θα γίνει στη Βόνη, Βόνη 23. Εμείς κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη και να δεσμευτούν για την χρηματοδότηση του σχεδίου του για την ισότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες, να υπάρχει χρονικό πλαίσιο, ε, ταξινόμηση προτεραιοτήτων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά αν θέλουμε να υπάρξει στήριξη στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία των Παρισίων. Είπαμε, η πρόκληση αυτή της κλιματικής αλλαγής θα γίνει όλο και μεγαλύτερη στο μέλλον. Κάτι άλλο ξεκάθαρο για μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν το κάνει. Δεν ε, σέβεται απόλυτα τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει σε διεθνείς συμφωνίες. Αν δούμε το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις ε, υψηλές θέσεις απασχόλησης, βλέπουμε ότι δεν το κάνει, ούτε και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερα, να αναλάβει πρωτοβουλία, να αναπτύξει ένα σύστημα επικοινωνίας όσον αφορά το θέμα αυτό της ισότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η κλιματική δικαιοσύνη είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Έτσι ε, θα προχωρήσουμε σε πολιτικές προσαρμογής Άμβληση των ε, συνεπειών, των επιπτώσεων και ε, με προγράμματα που ήδη υπάρχουν αλλά και με νέα. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει βοηθώντας τον ΟΗΕ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία νομική βάση για την μετανάστευση η οποία απορρέει από την κλιματική αλλαγή. Ξέρω ότι ο ΙΕ δουλεύει πάνω σε αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μεγαλύτερη της κλιματικής αλλαγής. Αυτά έχω να πω προς το παρόν και περιμένω τα σχόλια των συναδέρφων και την συμβολή τους στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Άγκστρομ. Ποιος θέλει παρακαλώ το λόγο από τους κοιόδης ηγητές κανεί, Κυρία Πιετικάιναν, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ο ΕΛΚ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που πήρε πολύ στα σοβαρά το θέμα και ήδη έκανε μεγάλες προσπάθειες για να εκπονήσει το σχέδιο ψηφίσματος. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία. Το σημαντικό εδώ είναι η γνώση ε, και το θέμα των οργανώσεων των ε, γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη και πόσοι πόροι, πόσα κονδύλια δίνονται στο ΚΕΓΕ, στο Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών. Μπορείτε να μα δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία για τα κονδύλια και ποιο είναι ο ρόλο των γυναικών στην, στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και τι δυνατότητε χρηματοδότηση υπάρχουν. Επίση, πώ ε, επηρεάζουν οι κλιματικές αλλαγές στους άνδρες και πώς τις γυναίκες. Υπάρχουν διαφορές. Επίσης, ε, αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία ήδη. Ότι το 1% των πιο πλούσιων στον κόσμο ε, δεν περιλαμβάνει πολλές γυναίκες. Ε, επίσης, έχουμε μεγάλες μεγάλα ποσοστά πληθυσμού που μένουν σε πολύ ευάλωτες περιοχές με μεγάλη φτώχεια και με μεγάλο εργατικό φόρτο το 70% των ανθρώπων που, έχουν, που εργάζονται πολύ περισσότερο ζουν με λιγότερα από 70 δολάρια τη μέρα, η ευρώ τη μέρα και το μεγαλύτερο ρυθμό αυτού του πληθυσμού είναι οι γυναίκες. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει μεταξύ των αναπτυσσόμενων και λιγότερων αναπτυσσόμενων χωρών αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κλιματικές αλλαγές είναι αυτοί που υποφέρουν λιγότερο και εκείνοι που έχουν το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επηρεάζουν λιγότερο τις κλιματικές αλλαγές είναι αυτές που είναι ο κόσμος που επηρεάζεται κυρίως και δεινοπαθεί από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Είναι μεγάλη αδικία λοιπόν που προκύπτει από αυτά τα στατιστικά στοιχεία και θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της κλιματικής δικαιοσύνης. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μερίδιο των κονδυλίων και των ε, πόρων και των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα που διαφέρει, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το ποιοι μολύνουν και ποιοι πληρώνουν τα σπασμένα, που δυστυχώς δεν είναι ίδιοι. Επίσης, οι γυναίκες όχι μόνο ε, πλήττονται κυρίως από τις κλιματικές αλλαγές και υποφέρουν από αυτές, αλλά έχουν κρίσιμο ρόλο στην ε, καταπολέμηση, την ε, πρόληψη των κλιματικών αλλαγών, αρκεί να τους δώσουμε την ευκαιρία να συμβάλλουν όπως μπορούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διατροφή και οι επιλογές, οι καταναλωτικές επιλογές που κάνουν οι γυναίκες και στις αναπτυσσόμενες και στις αναπτυγμένες χώρες. Λοιπόν, δώσουμε δύναμη στις γυναίκες, να δυναμώσουμε στο να επιλέγουν το, τοπικά προϊόντα, υγιεινά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, τότε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα μειωθεί αισθητά. Κατά ένα τρίτο ίσως. Και μιλάμε για καθημερινές καταναλωτικές επιλογές και διατροφικές επιλογές. Πώς λοιπόν θα δυναμώσουμε τις γυναίκες ε, με κατάλληλους πόρους ώστε να κάνουν σωστές επιλογές που θα έχουν το χαμηλότερο ε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άλλο θέμα είναι η βιώσιμη χρήση των πόρων. Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματίες γυναίκες ε, τοπικά έχουν λιγότερους πόρους και παραγωγικούς και υπάρχει με μεγάλη αδική ό,τι αφορά την πρόσβαση στους πόρους ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών αν αποκατασταθεί τέτοια ισότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα είναι μικρότερο και το αποτέλεσμα πιο βιώσιμο. Αν όμως η νομοθεσία μας δεν επιτρέψει αυτή την δικαιοσύνη στην πρόσβαση, πάλι θα εξωθούνται οι γυναίκες ε, να εγκαταλείπουν ε, τις περιοχές τους, να, γιατί δεν θα έχουν πολλές επιχειρηματικές ε, δυνατότητες και διεξόδους κάτι που αποβαίνει εις βάρος και του κλίματος και της ανάπτυξης. Τέλος. Πώς θα ενισχύσουμε τις γυναίκες στις διαπραγματεύσεις, όπως κάναμε και για την πρόληψη των συγκρούσεων. Πώς θα τις ενδυναμώσουμε και στα θέματα τα κλιματικά. Νομίζω ότι μπορούμε να τις ενδυναμώσουμε σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, σε τοπικό, περιφερειακό, σε πολιτικές μας για τη συνοχή δηλαδή στην εφαρμογή τοπικών ε, πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, να συνεργαστούμε με γυναικείες οργανώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες για να ενισχύσουμε τις γυναίκες στη συμμετοχή της λήψης στη λήψη αποφάσεων και στι ε, παγκόσμιε διαπραγματεύσει για τι κλιματικέ αλλαγές και πάλι είναι πολύ χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν επιτέλους να στείλουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα χειρό μήνυμα ότι Στι διαπραγματευτικές μας ομάδες και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσετε μία ισορροπία μεταξύ των φύλων στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον και για το κλίμα. Αυτά εν ολίγη, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πιετικά. Είναι ο κύριο Μαχτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι σκιώδης συγκητής. Θα αντικαταστήσω εδώ τον, τον σκιώδη εισηγητρία που μου έδωσε το κείμενό τη. Οι Σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες ε, στενίζονται αυτή την άποψη. Καταρχήν ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την ε, αξιέπαινη προσπάθειά τη. Με βάση τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το 2045 κίνδυνο ε, μετατόπιση 145 εκατομμυρίων στον κόσμο λόγω της απερίμωσης είναι δεδομένος. Ενώ με βάση τη Διεθνή Οργάνωση για τη Μετανάστευση 200 εκατομμύρια θα είναι οι συνάνθρωποι μας που θα χρειαστεί να μετατοπιστούν, να αλλάξουν τόπο κατοικίας μέχρι το 2050 λόγω των κλιματικών αλλαγών. Η, εκθέση, η δράση της έκθεσης για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές και ο αντίκτυπό του στις γυναίκες βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και στηρίζουμε την υιοθέτηση μιας μεθόδου που θα λαμβάνει υπόψη τα θέματα φύλου στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την πλατφόρμα για την μετακίνηση πληθυσμών λόγω θεομηνιών φυσικών καταστροφών και την προστασία για την προστασία των ε, ατόμων κατά τις ε, διασυνοριακές μετακινήσεις σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή κλιματικών αλλαγών. Ο σεβασμός των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και του σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα φύλων και τη χειροφέτηση των γυναικών μας βρίσκει επίσης σύμφωνος. Εφαρμογή νέων ε, δικτών ανάλογα με το φύλλο και η λήψη υπόψη του στα σχέδια δράση για την ισότητα των φύλων. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στην ενίσχυση τις θέσεις της εισηγήτριας και το, αυτό θα κάνουμε και με τις τροπολογίες. Τώρα, ως προς τις τεχνικές πτυχές, θα θέλαμε να ενισχυθεί η έκθεση σε δύο σημεία. Σε ό,τι αφορά την πολιτική χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων στα πλαίσια της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Επίσης, να εξασφαλίσουμε ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, αλλά και στην εφαρμογή των πολιτικών και άλλων δράσεων επιτόπου. Ε, επί του πρακτικού, ε, θα επιμείνουμε στην ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να ενισχυθεί η αυτόνομη πρόσβαση των γυναικών στην ε, ιδιοκτησία και στις δράσεις και να προσθέσουμε την ε, πρόσβασή τους σε, σε, τεχνογνωσία. Επίσης, να αποφύγουμε άσκηση βίας βάρος των γυναικών κατά την μετακίνηση των πληθυσμών και να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του σε περίπτωση μετανάστευση Επίσης, ε, ε, διαπαιδαγώγηση σε θέματα σεξουαλικά και αναπαραγωγικής υγείας, να προβλέψουμε αντίστοιχα σχέδια δράσης και να εξασφαλίσουμε και τη σωστή τους χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Κύριος Εκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερματική Πιετικά, έναν την εισηγήτρια για την ε, έκθεσή της, την οποία και υποστηρίζω αμέριστα. Όλοι βέβαια θυγόμαστε από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο η κλιματική αλλαγή δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλλο, ούτε στο βορρό ούτε στο νότο. Σε πολλές κοινωνίες οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην ε, γη, την ιδιοκτησία, την εκπαίδευση σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυσανάλογα υψηλό, ε, υποφέρουν από τη φτώχεια. 70% των ανθρώπων που ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας είναι γυναίκες και είναι λιγότερο σε θέση να αντιδράσουν στα προβλήματα και της κλιματικής αλλαγής όπως στον Νότο έτσι και στο Βορρά γιατί και εκεί οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και δεν μπορούν να ε, αντεπεξέλθουν στις ψηλότερες τιμές στα τρόφιμα ή στα ενεργειακά προϊόντα. Και επιπλέον οι γυναίκες έχουν επιτοπλίστων και την ευθύνη τις ε, προμήθειες για την οικογένεια σε τροφή τροφίμων, ενέργειας, ύδατος. Στην αφρικανική γεωργική οικονομία παραδείγματι το μεγαλύτερο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό ε, των τροφίμων παρέχεται από τις γυναίκες όπως γενικότερα σε όλο τον κόσμο αλλά έχουν ε, τα μικρότερα ποσοστά ιδιοκτησίας της αρρώσιμης γης περιοχή του Σαχέλ εντωμεταξύ λόγω της κλιματικής αλλαγής ε, εμφανίζει όλο και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας. Είναι πολλές φορές ανάγκη η γυναίκα και τα, κορίτσια, ε, και τα κορίτσι να περπατήσουν για χιλιόμετρα για να μπορέσουν να φέρουν νερό από όλο και πιο απομακρυσμένες πηγές. Ταυτόχρονα δεν έχουν συμμετοχή ή ε, δυνατότητα εκπαίδευση, δεν έχουν συμμετοχή στα κοινά, δεν έχουν πολιτικό λόγο. Έτσι λοιπόν Πρέπει να διαπιστωθεί ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την κατάσταση της υγείας των γυναικών και των κοριτσιών λόγω της θέσης του στην κοινωνία, ε, κατά κύριο λόγο και βέβαια λόγω και της έλλειψης ε, επαρκών τροφίμων. Οι εγκυμοσύνες οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν ιδιαίτερα κατά την περίοδο ε, της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεαστεί η γυναίκα και η υγεία της από το παράστο της ελονοσίας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό φαινόμενο. Ε, είναι λιγότερο καλά ενημερωμένε οι γυναίκε σε σχέση με του άντρε, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν και να προφυλάσσονται από του κινδύνου αυτού. Είναι θύματα τη κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα όμω οι γυναίκε έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό και ιδέε για την προστασία από τι κλιματικέ αλλαγέ. Έχουν ιδέε και δυνατότητε, τι οποίε σπάνια ε, υποστηρίζουμε ή διακυγνώσκουμε. Έχουν πολύ συχνά πολύ πιο οικολογική ε, στάση απέναντι στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Περπατάνε πιο περισσότερο από ό,τι παίρνουν το αυτοκίνητο, είπαν, ε, με το λεωφορείο, αντί για το ιδιωτικό μέσο μεταφοράς. Ε, τρώνε λιγότερο κρέας, είναι πολύ πιο οικολογικά συνειδητοποιημένες και στον ιδιωτικό τομέα. Ε, η διαχείριση από τον, τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους αλλά και της γενικότερης πολιτικής ξέρουμε ότι είναι στα χέρια των ανδρών και έτσι δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες και οι ιδέες των γυναικών σε τοπικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο Δυστυχώ πολύ σπάνια λοιπόν λαμβάνονται υπόψη οι ιδέε των γυναικών και όταν έχουμε αλλαγέ που προξενούνται από την κλιματική αλλαγή με συνέπεια τη μετανάστευση, πολύ συχνά οι γυναίκε μένουν ε, στην ε, πατρίδα του χωρί τα οικονομικά μέσα εκείνα ή τα, ο, τους πόρους που θα τους επιτρέψουν να στηρίξουν και να ε, θρέψουν την οικογένειά τους. Και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει ότι μέχρι το 2045 35 εκατομμύρια άνθρωποι στην υποσαχάρια Αφρική θα χρειαστεί να καταλήψουν τις συστήσεις τους και λόγω της επέκτασης της περιοχής της ε, ξηρής, της ερήμου. Κλιματολογική πολιτική λοιπόν χωρίς τη γυναίκα δεν είναι δυνατή. Πρέπει να αξιοποιηθεί το δυναμικό των ανδρών όσο και των γυναικών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, την υποστηρίξω πλήρω και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με την συνάδελφο ΣΕΠΑ. ΣΕΡΠΑ, ευχαριστώ. Η συγκεκριμένη πρέπει να φύγει δυστυχώς για το επόμενο θέμα για να πάει στην Επιτροπή Απασχόλησης. Γι' αυτό παρακαλώ Τώρα που έχουμε τρεις ομιλητές, να περιορίστε τις ομιλίες σας στο δυνατόν. Ξέρω ότι δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά μια και η κυρία Έγκστρομ θα πρέπει να φύγει. Είμαστε στο δυνατόν πιο σύντομοι, παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, η κυρία Ιούτο. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και συγχαρητήρια για αυτή την πολύ καλή βάση που έχει και τα θετικά στοιχεία περιλάβει, υπογραμμίζοντα σε παραδείγματα το γεγονό ότι οι γυναίκες είναι ναι μεν πιο ευάλωτες όσον αφορά τι κλιματικές αλλαγές, όλα αυτά που υπόθηκαν ήδη. Γιατί οι γυναίκες αυτές που έχουν λιγότερη πρόσβαση στους πόρους ή στην ε, εκπαίδευση, ε, στην εργασία ή έχουν λιγότερα ε, λιγότερε ευκαιρίε για διακτήσια ή εγγή και όλα αυτά. και ταυτόχρονα υπογραμτεί στην έκθεση ότι σε γη και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα υπογραμμίστε στην έκθεση ότι η Συμφωνία των Παρισίων λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι η αίσθηση του φύλου θα πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή τη υλοποίηση αυτή τη συμφωνία. Και επίσης ε, στην έκθεση καταγράφεται και η ιδέα της κλιματικής δικαιοσύνης, δηλαδή γίνεται η διασύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων και της ανάπτυξης και εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο ακόμα πτυχές που θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή αλλά ταυτόχρονα έχουν και ρόλο για πρόληψη της ε, κλιματικής αλλαγής στο πρώτο σημείο. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι γυναίκες έχουν ε, μεγάλες δυσκολίες και καταπλειονότητα δυσκολίες στις περιοχές που εμφανίζονται όλες τις φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για την πλημμύρα, είτε πρόκειται για την ξηρασία ή άλλες συνεπείς κλιματικές αλλαγής, ακριβώς γιατί αυτές είναι οι οποίες δουλεύουν τη γη, κάνουν αυτές τις δουλειές τις σχετικές με, με τον βασικό αυτό πόρο ο οποίος καταστρέφεται από την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα αυτές οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης που ακολουθεί τις κλιματικές ε, ε, καταστροφές. Χρειάζεται λοιπόν για τις γυναίκες να εξασφαλιστεί ε, υποστήριξη στην περιοχή όπου ζουν, στα εδάφευτα όπου διαμένουν και με τα βασικά αγαθά, νερό, τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη. Ταυτόχρονα βέβαια ο ρόλος της γυναίκας που όπως είπαμε μπορεί να έχει και προληπτική δράση για την κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί είναι πολύ πιο ευαίσθητες και ε, προσέχουν περισσότερο την κλιματική αλλαγή, έχουν ε, ε, συμπεριφορά που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στο κλίμα, στο περιβάλλον. Και γι' αυτό θα έπρεπε να συμμετέχουν και περισσότερο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων που θα επηρεάσουν ε, και θα προλάβουν αυτέ τι κλιματικέ αλλαγέ. Πρέπει λοιπόν να στηριχθούμε στην κατάρτιση, την συνειδητοποίηση και την ενδυνάμωση των γυναικών αυτών που θα μα βοηθήσουν για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. Ταντσίλα. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα σημαντική βρίσκω την πρόταση της εισηγήτριας για την έκθεση αυτή και συμμερίζομαι βεβαίως και τα λόγια της κυρίας Αγιούτο που μίλησε πριν από μένα αλλά και των λοιπόν συναδέλφων. είναι δεδομένο ότι στι ψηφοφορίε των περιπτώσεων οι γυναίκε είναι πολύ πιο ευάλωτε στην κλιματική αλλαγή, πολύ προστερό από του άνδρες είναι οι πιο φτωχές στον κόσμο, είναι πολύ πιο εξαρτημένες για την επιβίωσή τους από τους φυσικούς πόρους που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, μπορεί να αντιμετωπίζουν κοινωνικές, οικονομικές αλλά και πολιτικές δυσκολίες ή περιορισμούς που δεν τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν στις κλιματικές αλλαγές. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους λοιπόν για την επιβίωσή τους οι γυναίκες έχουν περιορισμένη κινητικότητα, περιορισμένη ή άνηση πρόσβαση στους φυσικούς σπόρους και γι' αυτό οι γυναίκες ιδιαίτερα στην Ήπεθρο πλήττονται δυσανάλογα βαριά από τις κλιματικές αλλαγές και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν και οι στρατηγικές σχετικές με το φύλλο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπογραμμίσουμε ότι οι γυναίκες δεν είναι απλώς ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να καταστούν και πρωταγωνίστριες στην ε, περιστολή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή. Έχουν ευρύτατες γνώσεις και εξειδίκευση που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη συγκράτηση των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών. Επίσης, έχουν την ευθύνη στις κοινωνίες τους αλλά και στις κοινότητες τις οποίες ζουν, διαχειριζόμενες τους οικιακούς αλλά και φυσικούς πόρους. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να, συνα... να συμμετάχουν, να να συμμετάσχουν ε, σε μια στρατηγική ζωής ε, πιο προσαρμοσμένη στην ε, περιβαλλοντική κατάσταση και τις κλιματικές αλλαγές. Ε, όταν προσδιορίζονται οι στρατηγικές για την ανάπτυξη και ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συμμετέχουν οι γυναίκες περισσότερο. Οι επικεφαλής αντιπροσωπιών γυναίκες, οι παραδείγματοι, ε, που εκπροσωπούν τα κράτη σε επίπεδο ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές, ε, είναι πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλότερη αυτή η συμμετοχή των γυναικών από ό,τι αυτή των ανδρών. Πρέπει λοιπόν να ενσωματωθεί και αυτή η διάσταση στο διάλογο για την κλιματική αλλαγή. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι υπάρχουν τέσσερις ε, τομείς πολύ σημαντικοί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής η συγκράτηση, η προσαρμογή, η μεταφορά τεχνογνωσίας και συνοδευτικά παρουσία ε, των γυναικών στην χρηματοδότηση. Εξασφάλιση για τις γυναίκες χρηματοδότησης ή της πρόσβασης, και της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και αυτό μπορεί να τις βοηθήσει να συμβάλλουν σε όλες αυτές ε, τις ε, σε όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μαρτζελέης είναι ο τελευταίος μου εδώ μιλητής στον κατάλογο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός γιατί θέλω να σας πω ότι έχουμε γραμμοδέτηση στη Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρία Σενέα. Είμαι εισηγητής υποφαινόμενος. Το παρουσιάσαμε την έκθεση την προηγούμενη Δευτέρα και ελπίζω να συγκεντρώσουμε μεγάλη πλειοψηφία και συνένεση σε όλα αυτά τα θέματα. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στις γυναίκες και στη διάσταση του φύλου στις χώρες του Νότου ε, και φυσικά και στον ενεργό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες ε, προκειμένου να κάνουμε τη μετάβαση σε ένα πιο καθαρό κόσμο και με λιγότερη ρήπαση. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι αυτή η δυναμική είναι απαραίτητη, γιατί θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στο γυναικό στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ε, γιατί ε, σίγουρα είναι, είμαστε εδώ πολύ λιγότεροι άνδρες, αλλά συνήθω ε, είναι πολύ περισσότεροι άνδρες που αποφασίζουν και θα πρέπει να έχουν και πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν παράγοντε αλλαγή οι γυναίκε. Επίσης, στην ε, στις πολιτικές ε, συνεργασίες και ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε και διάσταση φύλου μαζί με τη περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις φάσεις των σχεδίων, του σχεδιασμού, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τη διάρκεια και επίσης ε, σωστή συγκέντρωση στοιχείων και αναφύλλω. Γιατί θέλουμε μια πραγματικά καλά προσανατολισμένη αναπτυξιακή πολιτική που θα συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, χρειαζόμαστε τα ουσιώδη στοιχεία για να μπορέσουμε να δράσουμε. Άρα στοιχεία και αναφύλλω. Επίσης, ε, είναι σημαντικός ο ρόλος των γυναικών και στη Γεωργία, κυρίως στις χώρες του Νότου, που είναι ε, ε, ουσιαστικά γυναίκες αυτές που διατηρούν ε, τη διαβίωση των αισθειών ε, τους. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι επιπτώσει που έχουν οι φυσικέ εντό εισαγωγικών καταστροφέ, αλλά δεν είναι και πολύ φυσικέ γιατί η αιτία του που είναι οι κλιματικέ αλλαγές, είναι ανθρωπογενής παράγοντας. Και να δούμε τι επιπτώσει που έχουν οι φυσικέ καταστροφέ στι γυναίκε και πώ θα τι βοηθήσουμε για να προσαρμοστούν καλύτερα. Θα σα δώσουμε τη γνωμοδότηση αυτή και στην εισηγητρία φυσικά της έκθεσής σας, προκειμένου να τη λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Η προθεσμία για την ε, ε, υποβολή προτάσεων 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Στις 4 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια ε, θα ψηφίσουμε τον επόμενο Φεβρουάριο του 2018, δηλαδή στο Στρασβούργο. Πέραμε τώρα στο σημείο 6, την επόμενη έκθεση, την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σόιτροβα είναι η συγγετριά μας και θα της δώσω το λόγο για να μας κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση που δείξατε και θα ήθελα να σας κάνω την παρουσίαση του έγγραφου εργασία για τη διάσταση των φύλων, για την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ, που θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση της έκθεσής μου. Στο πρώτο τμήμα του σχεδίου, του σχεδίου εργασίας μιλούμε για τη σημασία που έχουν τα ΜΜΕ και τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι μόνο ένας ε, κλάδος, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο που επηρεάζει σημαντικά την κοινή γνώμη και τη διαμόρφωση κοινή γνώμη. Οπότε στόχο μου είναι να διαπιστώσω σε ποιο βαθμό εκπροσωπούνται επαρκώς οι γυναίκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη δημιουργία περιεχομένου, στη διαχείριση του περιεχομένου, αλλά και το πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τι γυναίκες. Θα υποδιαιρέσω την έκθεση σε διάφορα τμήματα. Καταρχήν, πεδίο εφαρμογή ε, και ορισμοί. Θα επικεντρωθούμε στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωση στον τύπο, ε, στα διαδικτυακά ε, δίκτυα. Δεν θα επεκταθούμε ιδιαίτερως γιατί δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Θα μιλήσουμε κυρίω για τα παραδοσιακά ΜΜΕ, τύπο και τηλεόραση. Επίση, θα αναλύσουμε το πώ παρουσιάζονται οι γυναίκε και πώ εκπροσωπούνται στα ΜΜΕ ω εργοδότε, εργαζόμενε και δημιουργοί. Επίση χρησιμοποιούμε διάφορε βάσει δεδομένων, το Eurostat, το, την πολυμορφία των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ευρώπη και το καθεξή. Έχουμε πολύ περισσότερε γυναίκε που αποφυτούν από δημοσιογραφικέ σχολέ, 68%. Επίση οι γυναίκε είναι σημαντική εργατική δύναμη αλλά υποεκπροσωπούνται σε επίπεδο διαχείρισης και στις θέσεις των ανώτατων στελεχών. Μόνο 8% των διευθυντών είναι γυναίκες. Δεν είναι αρκετή εκπροσώπηση. Επίσης, αναλύουμε τις φυστάμενες πολιτικές ισότητας και πρακτικές. Έχουμε πολιτική για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι ειδική πολιτική για την ισότητα φύλων στα ΜΜΕ. Επίσης, το βασικό νομικό μέσο είναι η τρίτη οδηγία για τα οπτικοκουστικά μέσα, που όμως δεν έχει καμία αναφορά της εκπροσώπησης των ανδρών και γυναικών στη διαδικασία, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, στα, στους ρυθμιστικούς φορείς. Θεωρώ ότι το περιεχόμενο μη ε, ε ε, δεν θα πρέπει να ρυθμίσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να προβάλλουμε καλά παραδείγματα και πρακτικές για την καταπολέμηση της φαλοκρατίας και του σεξισμού. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγετικές, ηθήνουσες και επίσης ε, θα εξετάσουμε και το ευρωπαϊκό αλλά και το εθνικό επίπεδο. Θα υποβάλω την, το σχέδιο έκθεσης μου ανάλογα με τα πορίσματα που θα συγκεντρώσω κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα Νοεμβρίου και περιμένουμε από ανυπομονησία τις προτάσεις και τις α, παρατηρήσεις σας. Ποιος θέλει το λόγο, εγώ είμαι σοσιαλιστές και όδηση, η Τζούλη. Τότε επιτρέψτε μου να πω εγώ δύο λόγια ως από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για ένα θέμα που συζητάμε στην Επιτροπή μας εδώ και χρόνια και εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Ακόμα, όπως είπατε, δεν υπάρχουν αρκετά, αρκετές γυναίκες στα υψηλά επίπεδα λήψης αποφάσεων στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό ισχύει σε όλες σχεδόν τις χώρες μέλη. Και είναι όλο και πιο δύσκολο να λυθεί αυτό. μιλήσαμε ήδη το 95 από το Πεκίνο όπου αναγνωρίστηκε ότι η σχέση των γυναικών με τα μέσα ενημέρωσης είναι κάτι πολύ σημαντικό για να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και εκεί μιλούσαμε για στόχους, στρατηγικές και προγράμματα δράσης. Χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή λοιπόν και πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων στα μέσα ενημέρωσης και στις τεχνολογίες τις ψηφιακές. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Και σήμερα υπάρχουν κάποια συμπεράσματα. Το έγγραφο αναφέρει διάφορα σημαντικά στοιχεία για τα καθήκοντα και τους ρόλους των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Λίγες όμως γυναίκες είναι εμπειρογνώμονες σε αυτό το κλάδο. Και όμως θα έπρεπε, γιατί μερικές φορές όταν κάποιος καλείται εμπειρογνώμων, δεν λέω πάντα, αλλά πολλές φορές ε, αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας λοιπόν έχει προβεί σε έρευνες πρόσφατα για αυτό το θέμα και στο 17% των περιπτώσεων, στα μέσα δηλαδή, οι γυναίκες θεωρούνται εμπειρογνώμονες. Δηλαδή ως επιτοπλίστων δεν θεωρούνται εμπειρογνώμονες οι γυναίκες, δεν θεωρούνται ειδικοί. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί όλο και περισσότερες είναι οι γυναίκες οι οποίες γνωρίζουν το θέμα τους, αλλά δεν αναγνωρίζεται αυτό. Δεν προσδιορίζονται ως ειδικοί. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Επίσης, στα μέσα ενημέρωσης γενικά εμποδίζονται οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε υψηλές θέσεις. όπως ε, συμβαίνει και σε άλλα επαγγέλματα, ναι μεν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά οι γυναίκες αυτές μένουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία, στη καινοτομία τους στα μέσα ενημέρωσης. Είτε πρόκειται για τα οπτικοακουστικά, δημοσιογραφία κλπ. Είναι σημαντικό. Δυστυχώς δεν βελτιώνεται. Μάλλον επιδεινώνεται η κατάσταση. Τώρα, αυτό το οποίο όμως δεν αναφέρει η έκθεση είναι τα, δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα. Και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εκεί πολλές φορές παρενοχλούνται κανονικότατα. Πρέπει να μας απασχολήσει αυτό γιατί τα κοινωνικά δίκτυα, facebook κλπ. αποτελούν όλο και περισσότερα μέσα επικοινωνίας. Γι' αυτό και πρέπει να τους δώσουμε σημασία, να δώσουμε σημασία στα τρόλς σε βάρος των γυναικών, στις επιθέσεις σε βάρος των γυναικών. Είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί και να βρεθούν οι κατάλληλες στρατηγικές να τα αντιμετωπίσουμε. Στον Ηνωμένο Βασίλειο έχω συνάδελφο που το έχει αντιμετωπίσει αυτό στο Twitter και βγήκε τελικά από το Twitter ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν πολλά είναι εδώ τα ζητήματα και είναι σημαντικά γιατί τα μέσα ενημέρωση είτε μας κάνουν είτε δεν μα κάνουν αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τις γυναίκες. Γι' αυτό πολύ χαίρομαι που υπάρχει έκθεση αυτή της εισηγήτριας και την ευχαριστώ και καλό θα ήταν η Επιτροπή μα να πάρει το θέμα σοβαρά και να το προωθήσει. Ευχαριστώ. Τώρα, ποιο. Α, η Τζούλη, η Τζούλη Βόρτ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι εδώ για τη Χάρη Χάρμαν που ήταν επικεφαλής ε, σε μέρος των Λέμπορ στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτιαξε μια επιτροπή γυναικών εκεί ακριβώς επειδή έγιναν αυτά που έγιναν με την Μύριο Ράιλι που ήταν ε, στο BBC, reporter δηλαδή, για ένα πρόγραμμα που ονομαζόταν Country File και συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα γιατί ήταν μεγάλη στην ηλικία και αυτό που μαζί τη παρουσίασε το πρόγραμμα, αλλά ήταν μεγαλύτερο από αυτήν στην ηλικία, αυτό συνέχισε να παρουσιάζει το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν οι διακρίσει είναι πολλαπλέ στον τομέα των μέσων ενημέρωση. Δεν είναι μόνο το ότι είναι οι είναι και το θέμα τη ηλικία. Η Χάρη να έκανε μια τεράστια εκστρατεία για να υποστηρίξει ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες στις ηλικίες μου για παράδειγμα έχουν να προσφέρουν πράγματα. Βέβαια ο Τραμπ έχει μια εκστρατεία κατά των γυναικών, το ξέρουμε αυτό, ε, να καταστέλλεται η φωνή των γυναικών, κάτι το οποίο βρίσκω πάρα πολύ σοβαρό. Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με την Τζιν Είναι μια οργάνωση στο κουρδικό Τουχιστάν που εξετάζανε το θέμα αυτό το σε βάρος των γυναικών, οι γυναίκες που είναι εκεί εξακολουθούν να κάνουν τους ρεπόρτες, να μεταφέρουν δηλαδή τα νέα από εκεί προς τον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια υπήρξαν ε, επιθέσεις προκειμένου να τις κάνουν να σοπάσουν. Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας και να υπερασπιζόμαστε τις γυναίκες αυτές που προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Γιατί ο κόσμος προσπαθεί να κάνει το αντίθετο με αυτές, να τις κάνει να σοπάσουν. Όταν έχουμε ανταποκρίτριες και τέντι στη χώρα μου για παράδειγμα και άλλες υπάρχουν καταπληκτικές γυναίκες που κάνουν μια δουλειά που θεωρείται στα μέσα ενημέρωσης ότι είναι δουλειά αντρών να είναι reporters δηλαδή σε δύσκολες περιοχές. Τα ονόματα των γυναικών reporters δεν ακούγονται καν. Εμείς πρέπει όμως να τους δίνουμε θέση στην κοινωνία μας και λόγο. Έπειτα, ε, γυναίκες που δουλεύουν ε, σε σταθμούς μπορεί να είναι γνωστά πρόσωπα, γιατί βλέπουμε το πρόσωπό του στο γυαλί όταν είναι στην τηλεόραση, όμως δεν τους δίνουν την ευκαιρία να συμμετέχουν επαρκώς στην ε, εκπόνηση του δελτίου ή στο περιεχόμενο των προγραμμάτων που παρουσιάζουν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Έκιο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Συγγετρία, σας ευχαριστώ για το πλήρωσα έγγραφο εργασία και ιδιαίτερα για τις στατιστικές που αναφέρεται σε αυτό, που ρίχνουν φως στο πρόβλημα. 17% των εργαζομένων στο χώρο των έντυπων μέσων ενημέρωση, είναι γυναίκες ε, με μεγάλα ποσοστά συνδεύξεων που παίρνουν από άντρες. Ε, υπάρχουν μελέτες ε, από πανεπιστήμια σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς ε, της ενημέρωσης που δείχνουν, δυστυχώς και αφορά τη Γερμανία αυτό, ότι οι γυναίκες έχουν υποεκπροσώπηση και στην τηλεόραση αλλά και στην παραγωγή την κινηματογραφική της Γερμανίας. Δύο άντρες πρωταγωνιστές αντιστοιχούν σε μία γυναίκα σε κύριο ρόλο. Επίσης ε, στις ενημερωτικές εκπομπές είναι υποεκπροσωπούμενες οι γυναίκες, 72% οι άντρες. 79% είναι οι ειδικοί που προσκαλούνται. Το ίδιο και στα quiz ή τα ε, reality shows. Πάλι κατά 80% τα παρουσιάζουν άντρες. Οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες ηλικία που μετράει από τα 30 χρόνια και μετά ε, μπαίνουν στο περιθώριο στην παραγωγή των ταινιών της τηλεόρασης αλλά και στην παρουσίαση των εκπομπών στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές, στις, ε, κινηματογραφ... στις κινηματογραφικές ε, Αυτό δεν συμβαίνει για λόγους τυχαία, ως διότι την σύμβαση, την, τις όρους της σύμβασης προσχωρήσουν οι άντρες οι οποίοι έχουν ως εκ τούτου απόλυτη εξουσία και για το κοινό στο οποίο θα απευθύνονται αυτές ε, οι εκπομπές ή οι ταινίες. Άρα μπορεί να παίρνουν ακόμη και πολιτικές αποφάσεις. Μπορεί αυτό να κρυθεί ως μια πολιτική απόφαση. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο πρέπει να εξεταστεί και υπό την πολιτική του πτυχή, όχι μόνο ως κοινωνικό πρόβλημα. Μία από τις συστάσεις που μας εξαγγέλει η συγγετρία ο ρόλος, παραδείγματι, της ε, ε, παρακολούθησης της τηλεθέασης και σε, με δείκτες πιο αναλυτικούς, νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικός, ε, σημαντική σύσταση. Επίσης χρειάζεται πιστεύω ένα παιδευτικός ρόλος της τηλεόρασης. Χρειάζονται σαφείς κανόνες, χωρίς οποίους δεν φαίνεται να λειτουργεί το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και επίσης, κοίταξα, ε, σε σχέση με τις Βρυξέλλες, πόσα ανταποκρίτριες γυναίκες υπάρχουν, ανταποκρίτριες των ιδιωτικών μέσων. Ε, το Spiegel, η Deutsche η Bild και άλλες εφημερίδες έχουν ε, από 28 ανταποκριτές, τέσσερις μόνο γυναίκες. Είναι μεγάλη ανισότητα. Και άρα πιστεύω ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια υποχρεωτική ποσόστοση. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ θέλει το λόγο. Ο κύριος Μαρτσελέση. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον στην εισηγήτρια για το έγγραφο εργασίας που υπέβαλε. Είναι σημαντικό αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες και προλαλήσασες για το ρόλο των γυναικών κυρίως στην εκπροσώπησή τους στις διάφορες σφαίρες λήψης αποφάσεων. Και εμείς οι πράσινοι θα θέλαμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του περιεχομένου, γιατί το περιεχόμενο είναι που προβάλλει μία πολύ ε, τυποποιημένη ε, εικόνα για τις γυναίκες, δηλαδή διονύζει αυτά τα στερεότυπα που Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι ο ρόλο και η εκπροσώπηση των γυναικών στα μέσα μαζική ενημέρωση. Κάτι που προποθέτει, όπω θα πει και η φαντάζομαι, ε, στην έκθεσή τη, ε, να επιμείνει πολύ περισσότερο στο θέμα αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει κάποιο ρόλο, να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε ε, μία εκδήλωση για τις ε, φαλοκρατικές διαφημίσεις και συνεργαστήκαμε με πολλούς δήμους και κοινότητες που προσπαθούν σε τοπικό επίπεδο να πατάξουν τις ε, διακρίσεις βάρος των γυναικών και μία φαλοκρατική παρουσίαση των γυναικών στις διαφημίσεις και ζητούσαν κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία οδηγία για τα θέματα αυτά, για παράδειγμα, το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες στις διαφημίσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να επικεντρωθούμε στην καλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διαμόρφωση του περιεχομένου και να δούμε πώς εκπροσωπούνται ώστε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, τα κλισέ και να ασχοληθούμε με θέματα συναφή με την φαλοκρατική παρουσίασή τους στις διαφημίσεις, στις εξιστικές διαφημίσεις. Ευχαριστώ. Δυστυχώ η συγκεκριά μα, η κυρία Σόιντροβα, χρειάστηκε να αποχωρήσει. Καταρχήν να πούμε τι βασικέ ημερομηνίε. Έκθεση του σχεδίου έκθεση προβλέπεται για τι 21 Νοεμβρίου. Και θα επιβεβαιώσουμε τις υπόλοιπες ημερομηνίε ημερομηνίες στις 21 Νοεμβρίου που θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και την προετοιμασία τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΛΤΑΠ μετά το 2020. Η συγκίτρια είναι κανονικά η κυρία Γκαρσία Πέρε, αλλά δυστυχώ κολλείεται σήμερα. Οπότε έστειλε την κυρία Ινέσα Αγιάλα Σέντερ που έχει την καλοσύνη να διαβάσει τη δήλωση τη εισηγήτριά μα κυρίας Πέρας. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντω με τιμά ιδιαίτερα αυτή η ανάθεση. Είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση στη χώρα και φανταστείτε τόσο περίπλοκη που χρειάστηκε η επικεφαλής αντιπροσωπεία μας να παραμείνει στην Ισπανία και με επιφόρτησε με την παρουσίαση της έκθεσης της, της γνωμοδότησης της μάλλον στο σχέδιο γνωμοδότησης που θα υποβάλλεται στην Επιτροπή προπολογισμών ε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η προετοιμασία τη ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, αυτή η θέση είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό η Επιτροπή σας θα πρέπει να προβάλλει τη, και να διατρανώνει τη θέση μας υπέρ της ισότητας των φύλων, την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και στον προϋπολογισμό, ώστε να ε, επικεντρωθούμε σε κάποια εγκάρσια σημεία και να διαμορφώσουμε ένα προϋπολογισμό που θα συνεκτιμά και τη διάσταση του φύλου και μάλιστα ως προτεραιότητα ε, σε όλα τα τμήματα του προϋπολογισμού. Σε μερικές περιπτώσεις, ε, σε μερικούς τομείς θα πρέπει να ανακτήσουμε τις, στο πρόγραμμα Δάφνη το το πρόγραμμα για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ηθαγένεια. Επίσης, θέλουμε κατάλληλο προπολογισμό, διαθέσιμη χρηματοδότηση που θα είναι εφάμιλη των, της φιλοδοξίας μας και της τεράστιας πρόσκλησης που δημιουργεί η καταπολέμηση της βίας της βάρος των γυναικών και της βίας λόγω φύλου. Και να καλύψουμε φυσικά και το θέμα της παιδικής ηλικία και να βελτιώσουμε τον προϋπολογισμό που είναι μειωμένος ε, στην πρόταση που έχει γίνει θα πρέπει να τον επαναφέρουμε στα προηγούμενα επίπεδα δεδομένων των τεράστιων αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω και της κρίσης αλλά και άλλων ε, πιέσεων στις οικογένειες και στην κατάσταση των γυναικών και στην εργασία, στο χώρο εργασίας και αλλού. Τις τελευταίες μέρες ε, είχαμε την παρενόχληση και τη βία ε, ακόμη και στο Hollywood, ένα θέμα που ε, βρέθηκε στη στο επίκεντρο της προσοχής των ΜΕ, θα πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ πιο φιλόδοξο τρόπο να καταπολεμήσουμε αυτή την βία εις βάρος των γυναικών, όποια μορφή και αν έχει. Επίσης, θέλουμε να αναφέρεται ρητά στον τομέα 3 της ασφάλειας και το, της ηθαγένειας ή προσημείωση κονδυλίων για την ισότητα των φύλων. Επίσης θα πρέπει να ανανεώσουμε την διοργανική μας δέσμευση υπέρ της δημοσιονομικής φιλοδοξίας, υπέρ του θέματος της ισότητας των φύλων. Στον τομέα 3 και επίσης ε, ζητούμε καλύτερη χρηματοδότηση μετά το 2020 και καλύτερη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό και γιατί όχι μια χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Δάφνη προκειμένου να προβληθεί καλύτερα και σε καμία περίπτωση να μην συρρικρωθεί και πάλι, να μην περικοπεί το συγκεκριμένο δημοσιονομικό κονδύλιο αν έχουμε ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού για το Δάφνη, θα εξασφαλίσουμε ε, την ακαιρεότητά του και την αποφυγή οποιασδήποτε απόπειρα περικοπή των σχετικών κονδύλιων στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά, αν έχετε απορίε, πολύ ευχαρίστω. Αλλά να τονίσω την υποχρέωση που έχει η Επιτροπή μα να αναγνωριστούν σε δημοσιονομικό επίπεδο αυτά τα θέματα τη ισότητα των φύλων για να αποσοβηθούν ε, οι γνωστοί κίνδυνοι και κυρίως να μην συρρυκνωθεί σε θέματα ισότητας ε, των φύλων ε, ο προϋπολογισμός. Γιατί οι ανάγκες όχι μόνο έχουν μειωθεί, έχουν αυξηθεί, οπότε τα αντίστοιχα κονδύλια θα πρέπει να περικοπούν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Σόνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου ε, των Πρασίνων θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της για αυτή την πρώτη εκδοχή της γνωμοδότησης και να πω ότι συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις που κάνει στο κείμενό της. Θα αποτελέσουν πολύ καλή βάση για την ε, θέση την οποία τελικά θα υιοθετήσει η Επιτροπή μας. Όσον αφορά τώρα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε πιο συγκεκριμένο το είδος Ευρώπης που θέλουμε για τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω πώς, εν περιπτώσει, έχουμε την ευκαιρία να πάμε πέρα από τις συζητήσεις, από τα σενάρια, από τις θεωρίες, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στις πολιτικές που χρειαζόμαστε, με συγκεκριμένα κονδύλια, με συγκεκριμένα προγράμματα προκειμένου να υλοποιηθούν. με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο βλέπουμε ποια Ευρώπη τελικά θέλουμε για τα επόμενα χρόνια. Και στον τομέα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων πολλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Τώρα συγκεκριμένα για τη γνωμοδότηση. Όσον αφορά την μεθοδολογία, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει προϋπολογισμός για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και να υπάρξει και μια πιο αυστηρή εφαρμογή που να συμπεριλαμβάνει πάντα την ε, διάσταση του φύλου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή πρόταση. Να συνεκτιμάτε πάντα διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορεί έτσι να μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην ισότητα από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα. Η ανακοίνωση τώρα της Επιτροπής για την αξιολόγηση δεν αναφέρεται στην εγκάρσια διάσταση του ζητήματος, κάτι το οποίο πιστεύω ότι αποτελεί αδυναμία στην υλοποίηση. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, προγράμματα κτλ. Συμφωνώ να αναφέρεται ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε ένα από τα κεφάλαια του επόμενου πολιτου δημοσιονομικού πλαισίου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ζωτική σημασίας για την εφαρμογή της διάστασης του φύλου εγκάρσια παντού σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο σε κάποιους τομείς, σε κάποια κεφάλαια, αλλά χρειαζόμαστε και ειδικά προγράμματα, κατάλληλα χρηματοδοτημένα βέβαια, για να πετύχουμε τον εγκάρσιο αυτό στόχο που είναι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Επίσης, η συγγήτρια λέει πόσο σημαντική είναι η επαρκής πρικοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία, το Δάφνη. Δυστυχώς ο προπολογισμό του προγράμματος Δάφνη μειώθηκε και τελευταία δεν έχουμε καν κονδύλι στον προπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως πρέπει να φροντίσει γιατί είναι αυτό που ελέγχει τον προπολογισμό. Οπότε να ζητήσουμε να ανακτηθούν αυτά τα κονδύλια και να βελτιωθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο. Θα υποβάλουμε τροπολογίες προκειμένου να προσπαθήσουμε, αν γίνεται να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την γνωμοδότηση αυτή. Θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες για να βελτιωθεί η υλοποίηση των στόχων υπέρ της ισότητας στον προπολογισμό και για την ενίσχυση των κονδυλίων που αφιερώνονται σε θέματα ισότητας και το Ταμείο Ισοτικών Επενδύσεων και το Δάφνη βέβαια. Και να φροντίσουμε να βρεθούν και άλλα κονδύλια. Το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κλέρ. Ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πιστεύω κι εγώ πως ναι, φυσικά και υπάρχουν έρητα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και μας απασχολεί πάρα πολύ όντως η χρηματοδότηση του προγράμματος Δάφνη. Πρέπει να διασφαλιστεί να υπάρξει συγκεκριμένη γραμμή και συγκεκριμένο κονδύλι. Όμως με απασχολεί και κάτι άλλο. Η τάση που αναπτύσσεται, που εντάξει φροντίσαμε για τις γυναίκες, φτάνει, το κάναμε. Οι γυναίκες είναι μια χαρά. Ας φροντίσουμε για απλοποίηση, οπότε ας το βγάλουμε από την ημερήσια διάταξη το θέμα. Και αυτό είναι που με τρομάζει, γιατί η συνέπεια είναι ότι θα χάσουμε αυτή την εσωμάτωση της διάστασης του φίλου σε όλες μας τις πολιτικές όσο προχωράμε στις συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάθεση και κάτι που αναφέρεται και στην έκθεση είναι το τι γίνεται με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων. Έχουμε ζητήματα έτσι κι αλλιώς και για άλλα θέματα, πόσο μάλλον για τη διάσταση του φύλου. Πώς λαμβάνεται υπόψη στον προϋπολογισμό. Πρέπει επίσης να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Τα ευρωπαϊκά ταμεία συχνά είναι και τα μόνα τα οποία βοηθούν στις χώρες μέλη και προσπαθούν να προσμετρήσουν αποτελέσματα. Ένα καλό παράδειγμα είναι να δούμε τις γυναίκες στον ακαδημαϊκό χώρο και πόσο δύσκολο είναι να φτάσουν σε μεταπτυχιακές, ε, σε ντοκτορά, Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το ε, ένα το πρόγραμμα πλαίσιο όπου περιλαμβάνεται η συμμετοχή τους σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Με τέτοιες προσπάθειες μπορεί να υπάρχει διαφορά και σε αυτό πρέπει να βασιστούμε. Και όχι να αφήσουμε αυτή την τάση τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες σιγά σιγά να μπαίνουν στο περιθώριο γιατί θεωρείται ότι έχουμε ήδη καταφέρει πολλά. Ευχαριστούμε άλλους κανείς. Ε, είναι απαντήσεις. Ναι, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τα σχόλια των συναδέρφων. Γιατί είναι πολύ σωστά και ενισχύουν Η συζήτηση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο φυσικά και θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη. Εξού και πρέπει να φροντίσουμε να μην χάσουμε ό,τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Το λέω αυτό έχοντας και στο μυαλό μου το Horizon 2020. Είναι κάτι καλό και γι' αυτό και πρέπει αυτή τη στιγμή να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο όπου τόσες δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα και όπου αυτή η γυάλινη οροφή, πως τη λέμε, είναι πιο γερή από ποτέ, δυστυχώς, στον ακαδημαϊκό χώρο. Σίγουρα δεν πρέπει να βασιστούμε στα μέχρι τώρα επιτεύγματα, γιατί πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά. Και ακριβώς επειδή έχουμε πετύχει μέχρι, μέχρι τώρα μερικά πράγματα, ο αγώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος και για να τα διατηρήσουμε, αλλά και για να πετύχουμε περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε στα επίπεδα του προπολογισμού τι προγράμματα, τι προσπάθειες μπορούμε να ενισχύσουμε. Δεν θα είναι εύκολο. Και όντω κινδυνεύουμε να πέσουμε στην παγίδα στην οποία αναφερθήκατε. Δηλαδή ότι ε, εντάξει, αφού το έχουμε βάλει τώρα την ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου παντού, εντάξει, το κάνουμε, φτάνει, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα πιο συγκεκριμένο. Ε, όχι λοιπόν. Είμαι σίγουρη ότι η συγγήτρια, η Ράτσα θα συμφωνεί με τα σχόλια των συναδέρφων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ όλους. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 23 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Δεκέμβριο, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τον Φεβρουάριο, αλλά είναι προς επιβεβαίωση και στην Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα θα πάει το θέμα το Μάρτιο, αλλά είναι προς επιβεβαίωση. Αυτά, αυτό ήταν το τελευταίο θέμα που είχαμε στην σε διάταξη για σήμερα. Διάφορα, υπάρχει τίποτα στα διάφορα, όχι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε. Επόμενη συνεδρίαση, προσεχή συνεδρίαση τα γυαλιά μου, θα βλέπω λέει η Πρόεδρος, είναι η 6η Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Και τώρα έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών.